For... Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, διότι άργησα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε την ημερήσια διάταξη μπροστά σας. Είσαστε ικανοποιημένοι. Εάν ναι, μεταβαίνουμε στο επόμενο θέμα. την πολιτική ε, δαφικότητας. Κυρία Ρόσμπαχ, πρόγραμμα για το ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον και το μέλλον στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η κυρία ε, Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα πολύ σύντομο θέμα. Έχουμε τα μία συνοχής και η πολιτική συνοχής είναι μεγάλης ύψης της σημασίας. Εάν προέρχεται από μία μικρή περιφέρεια όπως εγώ, συνειδητοποιείτε πόσο είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Εάν δεν υπάρχει η σωστή υποδομή. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε όσοι διαβιούν εκτός μεγάλων πόλεων και αστικών κέντρων, σε πιο απομακρυσμένες δηλαδή περιφέρειες, να έχουν μια βιώσιμη πολιτική μεταφορών. Επειδή προέρχομαι από μια τέτοια περιοχή, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό η Επιτροπή να ε, δει πού υπάρχουν οι βέλτιστες πρακτικές και να τους προσδώσει μία συνοχή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την πολιτική μεταφορών και πολιτική χρηματοδότησης. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να αφήσουμε να αναθέσουμε στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξει αυτές τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε όλοι να ευεργετηθούν από αυτές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη, μεγαλύτερη σαφήνεια και περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα τα οποία ήδη εφαρμόζονται και να ενημερώνουμε τους ε, πολίτες και τα κράτη-μέλη για τις πολιτικές αυτές. Αυτό είναι και το κύριο μέλημά μου Βεβαίως έγινε λόγος και για ε, ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων και θα πρέπει να δώσουμε απτά παραδείγματα σε ολόκληρη την Ευρώπη για να δούμε πώς ε, λειτουργούν και οι συνδυασμένες μεταφορές. Θα πρέπει να διαθέτουμε αποτελεσματικά δίκτυα έτσι ώστε να μπορούμε να μεταβούμε από το σημείο Α στο Β στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταθούμε περισσότερο στους σιδηρόδρομους, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τις αδικές μεταφορές και να στραφούμε στις σιδηροδρομικές. Ο κύριος Ρικέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω και την κυρία Ροσμπάχ για τη δουλειά της και την ευχαριστώ επειδή η πρώτη παρατηρήση που θα κάνω είναι ότι μας λείπουν ε, έγγραφα. Δεν είναι διαθέσιμη η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής ακόμα και υπάρχουν ελάχιστα έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ λαμβάνουν χώρα για τη διακυβέρνηση σημαντικές συζητήσεις. Θα υπογράψω, υπογραμμίσω απλώς κάποια σημεία που μου φαίνονται σημαντικά σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας. Η πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι οι αστικές περιοχές συγκεντρώνουν τα περισσότερα προβλήματα των μεταφορών, προβλήματα συμφόρησης και ρήπανσης. Είναι λοιπόν αυτό κυρίως ένα πρόβλημα που οφείλεται στις μεταφορές, αυτή η συμφόρηση. Οι αστικές περιοχές, δεύτερη παρατήρηση, είναι κόμβοι, αποτελούν κόμβους κυκλοφοριακούς, διατροπικούς, μονοτροπικούς ή διατροπικούς κόμβους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη διασύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις με το υπόλοιπο δίκτυο. Η κατάσταση λοιπόν αυτή επηρεάζει το σύνο της ε, πολιτικής μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αστικές περιοχές αποτελούν 85% του ΑΕΠ και 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Οπότε η συνοχή σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους είναι ουσιαστικό στοιχείο πολιτικής και ε, επίσης σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι μεταφορές αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της συνοχής των αστικών περιοχών. Η αποτελεσματικότητα των μεταφορών αγαθών και εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές είναι επίσης ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και ένα περιβαλλοντικό διακύβευμα, διότι σε αυτές τις περιοχές τις αστικές ε, υπάρχουν τα σοβαρότερα προβλήματα συμφόρησης και ρήπανσης που αγγίζουν, που αφορούν ένα πολύ υψηλό αριθμό ανθρώπων. Τέλο, τα προβλήματα χρηματοδότηση και διακυβέρνηση. Συμφωνώ με αυτά μαζί, η κυρία Μπαχ ω προ την ανάγκη να θεωρήσουμε ότι η διακυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα ε, σε ε, εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της επικουρικότητας αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια καλύτερη χρήση, μια καλύτερη χρήση, αξιοποίηση των πόρων των ε, διαρθρωτικών ταμείων και προφανώς θα χρειαστεί να σκεφτούμε την διασύνδεση μεταξύ τοπικού και αστικού επίπεδου σε ό,τι αφορά τα θέματα της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαβίσα. Η κυρία Σαβίσα, λέει ο πρόεδρος μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Yes. Yes. It was sometimes Mr. Ε, ε, δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρόσμπαχ για τη δουλειά της. Εκ μέρους της ομάδας μου θα, θέλω να πω ότι θα κάνουμε κάποια σχόλια και κάποιες, θα καταθέσουμε και κάποιες τροπολογίες την Δετάρτη σχετικά με τα σημαντικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε η συγγήτρια και έτσι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Is Κρέιμερ. Κύριος ή κυρία Κρέιμερ. Ο κύριος Κρέιμερ. Δεν ξέρω ακριβώς, θα με βοηθήσετε εσείς, λέει ο κύριος Κρέιμερ. Also, Einmal auch äh, schönen Dank für die Vorlage. Ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση και για αυτά τα έγγραφα. Ε, γιατί μιλάμε για μειονεκτικές περιοχές στις πόλεις υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα για το μέλλον, αλλά και οι μεγαλύτερες δυνατότητες να αντιμετωπιστούν και να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα αφενός, αλλά υπάρχουν και τεράστιες δυνατότητες για την επίλυσή τους πώς θα είναι η πόλη στο 2050. Η κινητικότητα δεν θα έχει πλέον τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό δεν αρκεί να προωθήσουμε τις μεταφορές μόνο στις μειονεκτικές περιοχές, αλλά παντού. Πρέπει το αυτοκίνητο να αντικατασταθεί από άλλα πιο φιλικά προς το χρήστη μεταφορικά μέσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ε, κάποια περιορισμοί ταχύτητας, κάποια περιορισμοί ταχύτητας σε ορισμένους δρόμους. Δεν πρέπει κανείς να ξεπεράσει δηλαδή τα 30 χιλιόμετρα. Γιατί να μην ισχύει αυτό για το σύνολο των πόλεων, για, όλη, για ολόκληρη την πόλη. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα κινητικότητας και αηφορίας Στις δύο πρωτοβουλίες, ε, ε, υπάρχουν ε, οι σχετικές πρωτοβουλίες και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αηφόρο βιώσιμη κινητικότητα. Όλες οι πόλεις που χρηματοδοτούνται από την Ένωση θα πρέπει να, έχουν, να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα, να καταρτίζουν ένα σχέδιο αηφόρου βιώσιμης κινητικότητας και να αναζητούν και άλλες λύσεις και άλλες πηγές χρηματοδότησης και να μην στηρίζονται μόνο στα σπόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί τη συγχρηματοδότηση τώρα διατυπώσαμε μια πρόταση. 60% για το οδικό δίκτυο και τα υπόλοιπα για το σιδηρόδρομο και το ποδήλατο από τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Η απόφαση πρέπει ωστόσο να... Που, θα πάρει όμως την απόφαση για το αν θα κατασκευαστεί ένας ε, δρόμος, μια οδός ή ένας ποδηλατόδρομος στις πόλεις. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, όταν επενδύουμε τεράστια ποσά στο οδικό δίκτυο, δεν είναι σωστή η λύση αυτό. Πρέπει να προβλέψουμε και ένα σημαντικό ποσοστό για το, τις διαδρομικές μεταφορές και επίσης ένα σημαντικό ποσοστό για τους κατασκευή ποδηλατοδρόμων. Μέχρι το 2030, 70-75% να καλύπτει αυτά τα νέα έργα. Όπω 20 Όπως είναι η γέφυρα της Μεσίνης, παραδείγματος χάρη. Βεβαίω, αν εστιαστούμε στα μεγάλα έργα δεν θα υπάρχουν αρκετά κονδύλια για άλλα μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά έργα. Ναι, εμείς εκτιμούμε πλήρως την σχέση της κυρίας Ρόντμπαχ. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση μετριοπαθής και αυτό ιδιαίτερα εκτιμούμε διότι το κλίμα όταν πρόκειται για τις αστικές περιοχές εκεί είναι άλλες αρχές που είναι αρμόδιες και όχι αστικές αρχές και ευρωπαϊκές. Εκτιμώ ιδιαίτερα την δέσμευση που, της κυρίας Ρότσμπαχ και βρίσκω ότι είναι σημαντικό να επισύρει την προσοχή πάνω ε, στην κράτηση, την ολοκληρωμένη, στο σύστημα ολοκληρωμένης κράτησης εισιτηρίων. Τα βλέπω αυτά τώρα στην γνωμοδότηση της ε, κυρίας Ροσμπάχ και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, σκέφτομαι επίσης ε, η παράγραφος 8 του εγγράφου. Στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι ποιες είναι οι δυνατότητες του Ταμείου Συνοχής για το, την ολοκλήρωση του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Είναι μια σύζευξη, μια σύνδεση κάπως αποτυχημένη για μένα και ε, για μένα, για την ομάδα μου είναι σημαντικό τα διευρωπαϊκά δίκτυα να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στα δίκτυα της Ευρώπης και από την άλλη πλευρά υπάρχει το Ταμείο Συνοχής. Το Ταμείο Συνοχής έχει ως αντικείμενο να βοηθήσει τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης και η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις ζώνες ε, κλειδί και στις πτωχές ζώνες στα διευρωπαϊκά δίκτυα με το Ταμείο Συνοχής μου φαίνεται ότι η σχέση αυτή εδώ είναι αδύναμη. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε, να προσαρμόσουμε το κείμενο της παραγράφου 8. Και έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο. Ξέρετε ότι πάρα πολλές δημόσιες μεταφορές ανάμεσα στις αστικές περιοχές ε, υπάρχουν ε, κυρίως ε, με πλοία. Έχουμε στην Ολλανδία την σχέση ανάμεσα στις δημόσιες μεταφορές και στις αστικές ζώνες του Νότου. Υπάρχουν συνδέσεις πάρα πολύ σύντομες χάρη στους ποταμούς, στις πλωτές οδούς και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση κειμένου που να περιλαμβάνει αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ κύριε Ζέλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση ε, παρουσιάζεται στα πλαίσια της ε, περιφερειακής ανάπτυξης και όλα αυτά θα ενσωματωθούν στην πολιτική της συνοχής. Στη συζήτηση που έχουμε τώρα υπάρχει το θέμα των πόλεων, των αστικών περιοχών που θα πρέπει να ε, ενταχθούν περισσότερο στη μελλοντική πολιτική της συνοχής. Αυτή είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία ε, θα πρέπει να εστιαστεί αυτή η έκθεση. Ε, όταν μιλούμε για τα δίκτυα, για τις πολλαπλές μεταφορές, θα πρέπει να δούμε αν η κινητικότητα, η αστική οι αστικές μεταφορές θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη στρατηγική. Διότι εκεί τίθεται ε, το πρωταρχικό θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Οι πόλεις είναι ε, ζώνες όπου ζει το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Και το θέμα της αστικής κινητικότητας πρέπει να σταθμιστεί ευρύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Από ό,τι τώρα. Οι πολιτικές της συνοχής θα πρέπει να δώσουν τα κατάλληλα κίνητρα και ενθαρρύνσεις και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο στην έκθεση κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ κύριε Μπράτμπουρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω, ακούγοντας τον κύριο Κράμερ, ότι ε, κάποιος κωδικοποιήθηκαν οι σκέψεις μου ε, σε σχέση αν υπάρχουν κίνδυνοι ακολουθώντας αυτό το δρόμο. Βεβαίως συμφωνώ με την εισαγωγή της κυρίας Ροτμπαχ και με τον κύριο Βαντάλεν. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ κίνδυνος σύγχυσης ε, ποια είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής συνεχής ο κύριος Μακδόναλ και άλλοι πρότειναν και συμφωνώ ότι τα θέματα αυτά από την άποψη των μεταφορών σχετίζονται ή με τις εθνικές πολιτικές ή με τις τοπικές πολιτικές. Και εγώ δεν θα ήθελα εμείς να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο που προτείνει νομίζω ο κύριος Κράμερ να προσπαθούμε να υπαγορεύσουμε ποιε επενδύσεις θα πρέπει να πάνε στις αστικές περιοχές στον τομέα των μεταφορών. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέμα τοπικό, τοπικών αποφάσεων, εθνικών αποφάσεων. Και δεν έχω κανένα ε, πρόβλημα με την ε, πρόταση της κυρίας Ντρόντμπαχ για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Αλλά ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να διοχετεύσουμε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό των μεταφορών. Είναι ένα θέμα τοπικής και εθνικής αρμοδιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοβατσέκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας τους συναδέλφους μου, ε, σύμφωνο περίπου με όλα τα όσα ελέγχθηκαν εδώ, αλλά ένα πράγμα δεν είναι αρκετά σαφές ε, για μένα. Νομίζω ότι υπάρχει μια ειδική προσέγγιση που ζητείται για να τονιστεί η σημασία των δημοσίων μεταφορών ε, για τις περιοχές όπου υπάρχουν μειονεκτούντα άτομα, άτομα με ειδικέ ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι σημαντικές για κάθε σημαντική πόλη. Μπορεί μια πόλη να μειονεκτεί απλώς επειδή υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμιακή, διότι υπάρχουν συμφορήσεις ε, στην κυκλοφορία και οι δημόσιες μεταφορές θα μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις αυτές και που θα μπορούν να διανοίξουν το δρόμο για την κινητικότητα των μεταφορών. Αυτό θέλω να τονίσω, ιδαλλιώς συμφωνώ με τα όσα είπα, λέχθηκαν. Οι πόλεις είναι ε, χώροι κατοικίας όπου ε, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μετακινούνται εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το αστικό περιβάλλον και η αστική κινητικότητα είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα για την προσεχή περίοδο και ελπίζω ότι συζητώντας τη μελλοντική πολιτική συνοχής, η πολιτική για τις αστικές μεταφορές να κατέχει τη θέση που της ανήκει. Αυτό σας το λέω διότι οι περισσότεροι ρήποι παράγονται από το αστικό περιβάλλον και γι' αυτό θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις δημόσιες μεταφορές έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικές και πιο οικολογικές αυτές οι αστικές πολιτικές μείωσης των ρήπων. Επίσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια οδηγία ήδη έτσι ώστε οι δημόσιες μεταφορές να είναι όσο το δυνατόν πιο οικολογικού χαρακτήρα. Γι' αυτό οι δημόσιες αρχές όταν οργανώνουν τους διαγωνισμούς είτε για την αγορά λεωφορείων είτε για την ε, ενοικίασή τους να λαμβάνουν υπόψη το κόστος για όλη την διάρκεια χρήσης αυτού του οχήματος, καθώς και το κόστος που ενέχεται, που αφορά μάλλον, την εκπομπή ρήπων. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να εξεύρουμε ευφύ συστήματα μεταφορών, έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα και να εξασφαλίσουμε μία σωστή πολιτική αστικών μεταφορών. Όταν μιλάμε για αστική κινητικότητα, μιλάμε για ευάλωτες ομάδες, αλλά και για τις επενδύσεις στις ε, υποδομές ιδιαίτερα στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως ως προς την αστική κινητικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα κατάλληλα μέσα για τις επενδύσεις αυτές και να αρκεστούμε στην αρχή της επικουρικότητας, διότι όταν μιλάμε για αστική πολιτική μεταφορά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τοπικές αρχές έχουν τον πρώτο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή. Δεν θέλει να λάβει το λόγο. Πολύ ωραία. Κύριε Ροσμπαχ, έχετε κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε σε αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτά που είπαν και θα προσπαθήσω... Πρέπει να πω ότι πολλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην Ευρώπη υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα οργάνωσης των κοινωνιών μας. Από τη μια έχουμε το μεγαλύτερο, την, το μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμού που συγκεντρώνεται σε αστικά κέντρα, αλλά υπάρχουν και χώρες όπου δεν ισχύει αυτό, που έχουμε τον πληθυσμό που είναι μοιρασμένο σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό αυτό δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα στο ένα ή το άλλο σχήμα. Διότι εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου ο πληθυσμό είναι μοιρασμένο σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν κατοικίε παντού σε όλη τη χώρα. Η Φιλανδία, αντίθετα και άλλες χώρες, σε αυτές υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις οπου δεν κατοικεί κανείς. Και μετά μικρές κοινότητες, οι οποίες ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γι' αυτό δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε πόλεις αφενός και αγροτικές περιοχές αφετέρου. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ τις βέλτιστες πρακτικές. Διότι έχουμε δύο τελείως διαφορετικές δομές στις χώρες μας. Συμφωνώ ότι υπάρχει ρήπανση στις πόλεις, ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα, την ποιότητα και την καθαρότητα, την μείωση της ρήπανσης που προκαλούν τα μέσα μεταφορών. Αλλά υπάρχουν και ορισμένες χώρες όπου τα χρήματα πηγαίνουν αποκλειστικά στις πόλεις με αποτέλεσμα οι άλλες περιοχές να υποφέρουν και να κινδυνεύουν να πεθάνουν. Άνθρωποι που κατοικούν σε μικρότερες κοινότητες, σε αγροτικές περιοχές, έχουν περιορισμένες δυνατότητες για μάθηση, για να πάνε στο σχολείο, να σπουδάσουν. Τα υγειονομική περίθαλψη είναι ανεπαρκής κλπ. λοιπά. Γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε αυτές τις περιοχές αναζητώντας και πάλι τις βέλτιστες πρακτικές και να μην στρέψουμε όλη μας την περιοχή, να μην συγκεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες και όλη μας την περιοχή στις αστικές περιοχές. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου δεν είναι όλος ο πληθυσμός συγκεντρωμένος στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ευχαριστώ όλους για αυτά που είπαν. Πήρα πάρα πολλές σημειώσεις. Θα προσθέσω ορισμένα πράγματα στο κείμενο και προσβλέπω, προσβλέπω στις τροπολογίες που θα καταθέσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροσμπαχ. Ήταν για μένα τουλάχιστον πάρα πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπατε. 10 Νοεμβρίου τελική ημερομηνία κατάσταση τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στην 1η Δεκεμβρίου στην Επιτροπή και ψηφοφορία στην Επιτροπή την Περιφερειακή Επιτροπή θα γίνει τον επόμενο χρόνο, τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Λόγω του χρονοδιαγράμματος ε, της Περιφερειακής Επιτροπής. Έκθεση Κράμερ. Πολιτική ανταγωνισμού. Μάικλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τον θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ εκείνων που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση ώστε να υπάρξει ουσιαστικός πραγματικός ανταγωνισμός θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στις τροπολογίες 10 και 11. Περιβαλλοντικά κριτήρια, περιβαλλοντικοί κανόνες. χρειάζονται τέτοιοι κανόνες για θεμητό ανταγωνισμό, αν θέλουμε να, να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ορισμένες εγγύησεις. 15 και 16 Για αυτές τις τρεις τροπολογίες θα ήθελα να πω αν πρέπει να κάνουμε κάτι για τη διάκριση ανάμεσα στις ε, ε, σιδεροδρομικές μεταφορές και τις οδικές μεταφορές. δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Στη Σλοβακία έχουμε μια μεγάλη αγορά για τις υδροδρομικές μεταφορές χωρίς άλλες αναλλακτικές δυνατότητες προώθησης των οδικών μεταφορών, διότι υπήρχε ένα ανώτατο όριο. Γι' αυτό κατέθεσα αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία. Μόλις έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για την ψηφοφορία, για την τροπολογία 18, που ζητά να μην γίνει χωριστή ψηφοφορία. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή αντιλήφθηκε ότι ο φόρος για το τροχαίο υλικό είναι κάτι το δύσκολο μπορεί να εφαρμοστεί, διότι υπάρχουν προβλήματα στη Γαλλία, αντιρρήσεις αμφισβητείται αυτή η πρόταση, διότι ο φόρος ανταγωνισμού έχει ε, μειωθεί σημαντικά ε, στη Γαλλία και αποφασίστηκε η καταβολή ενός φόρου για το τροχαίο υλικό. Οι μεταφορικές εταιρείες της Γερμανίας, της Ολλανδίας, Ελβετίας υποχρεώνονται να εφαρμόσουν διπλή φορολογία εφόσον όταν, αν χρειαστεί να πληρώσουν αυτό τον φόρο για το τροχαίο υλικό. Αυτό αντιβαίνει στην έννοια του θεμητού ανταγωνισμού και ευτυχώς που αποσύρθηκε αυτή η πρόταση. Από 19 μέχρι 20, τροπολογίες 19-20, δεν μπορούμε να δεχθούμε στους σιδηροδρόμους. Αν υπάρχει μια καθυστέρηση μια ώρας, πρέπει να επιστραφεί το 25% του εισιτηρίου και κάτι περισσότερο και το ποσοστό αυξάνεται ανάλογα με την καθυστέρηση. Αν δούμε όμως τι γίνεται με τις αεροπορικές εταιρείες. Λέμε στους επιβάτες ότι θα καθυστέρησε η άφηξη του αεροσκάφους. Δεν θα έπρεπε και εκείνοι να αποζημιώνονται για αυτή την καθυστέρηση και τα σλότ και οι συνδέσεις καμιά φορά είναι, έχουν τόσο πολύ στενά χρονικά περιθώρια που είναι αδύνατο να αποφευθεί η καθυστέρηση. Και επειδή εξοικονομούν χρήματα, οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να ακολουθούν αυτό το σύστημα. Μιλήσαμε αρχή για, για, τους, για καθυστέρηση πέντε ώρων για την αποζημίωση των ε, επιβατών. Το μειώσαμε στις τρεις ώρες. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό πρέπει να ισχύουν παντού τα ίδια πράγματα. Είτε πέντε ώρες για όλους, είτε μία ώρα για όλους. Όλους τους επιβάτες, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις ανάμεσα στους σιδηροδρόμους και τις αεροπορικές μεταφορές. δίκαιη αποζημίωση και άλλες ενώ σε άλλες τροπολογίες χρησιμοποιείται άλλη ορολογία για θεμητό ισότιμο ανταγωνισμό. Και εγώ δεν συμφωνώ σε ορισμένες περιπτώσεις με, αυτές, με αυτή τη διαφορετική διατύπωση. Τροπολογία 26 Εδώ θέλουμε, ζητάνε να διαγραφεί η λέξη dumping. Υπάρχουν πρακτικές dumping που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Πρέπει να βελτιώσουμε μέσα, μέσα, μέσα από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τον ανταγωνισμό, ώστε να προσφέρουν οι εταιρείε καλύτερες υπηρεσίες που θα προσελκύουν περισσότερους πελάτες. 26 έως 28. Δεν συμφωνώ με αυτές τις τροπολογίες. Και μετά έχουμε τρεις συμβιβασμούς, τρεις συμβαστικές λύσεις. Η πρώτη, α. Έχουμε τρεις τροπολογίες που καλύπτουν τα πάντα και το αποτέλεσμα με ικανοποιεί και γι' αυτό τις υποστηρίζω. Συμβιβασμός β εσωτερικές συνδέσεις. Και πάλι εδώ είναι θέμα ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας και πώς συμφιλιώνονται αυτά τα δύο, αυτές οι δύο έννοιες. Μπορεί να ισχύει για μεγάλες εταιρείες, αλλά βγάζουμε από την αγορά τις μικρές εταιρείες. Οι μικρές εταιρείες είναι οι πιο καινοτόμες και πρέπει να τους δοθούν κατάλληλες ευκαιρίες. Πρέπει λοιπόν να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες εταιρείες ανάμεσα στην, θέλουμε να προωθήσουμε ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα και για τις μικρές και για τις μεγάλες εταιρείες. Και είχαμε το, και ετέθηκε το θέμα για τα πόσο θα πρέπει να περιλάβουμε όχι τον τουρισμό, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το δεχθώ. Ο κύριος Μπαχ, Έλκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αγαστή συνεργασία την οποία είχαμε και από την οποία επωφεληθήκαμε. Δεν μπορεί να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός χωρίς κανόνες, αλλά θα πρέπει να εκπονηθούν βεβαίως αυτοί οι κανόνες και θα πρέπει να, ε, να έχουν απαιτήσει τακτικές. Αρχίζοντας θα ήθελα να πω ότι με όλη την εργασία την οποία έγινε η πρόταση αυτή είναι ικανοποιητική. Μπορεί βεβαίως ε, να εστιάσει κανείς την προσοχή στο 2009 ε, και να δούμε μια προοπτική για τις ε, επόμενα χρόνια για να δούμε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τον τουρισμό, έχουμε τις απαιτήσει από την Κομισιόν. Το ίδιο ισχύει και για τους διάφορους φόρους και εισφορές. Και η τροπολογία για ε, τα διάφορα δεν πρέπει να αρχίσουμε ε, μια τέτοια διαδικασία. Η Επιτροπή, όπως λέχτηκε, θα αναλάβει πρωτοβουλία στους τομείς αυτούς σε πολλές τροπολογίες το θέμα του ανταγωνισμού μόνο, όχι μόνο μέσα σε ένα μέσο μεταφορικό, αλλά ανάμεσα στα μεταφορικά μέσα και μέσα σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή η μορφή ελέγχου, αυτή η μορφή φορολόγησης είναι η κατάλληλη. Ο εισηγητής δεν χαιρέτησε την διαγραφή της τροπολογίας 10. Η ομάδα μας δεν ήθελε να διαγραφεί. Θέλουμε να έχουμε μια διάκριση ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών και στην ασφάλεια και στα κοινωνικά στοιχεία. Χαιρετίζω το όσα έγιναν με την τροπολογία για το dumping. πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό. Νομίζω ότι ε, γενικά είμαι υπέρ ε, της γνωμοδότης. Ευχαριστώ ε, κυρία Τίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κράμερ για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και με τους σκιώδεις και με σκοπό να φτάσει σε αυτές τις προτάσεις. Όταν μιλάμε για τον ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πληρούμε τις υποχρεώσεις της εσωτερικής αγοράς και αν όχι, ποια είναι τα εμπόδια. Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας, ο τομέας των μεταφορών συνδέει αυτό το κομβικό στοιχείο και με άλλους τομείς, διότι η απασχόληση εκατομμύρια θέσεων εξαρτώνται από την απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται και από την ανταγωνιστικότητα και από το πώς την διασφαλίζουμε στον τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό προσπάθησα μέσω ορισμένων τροπολογιών να ενισχύσουμε την ε, υπόθεση της σωστής, της υγιούς ανταγωνιστικότητας, έτσι ώστε να άρθουν και τα προσκόμματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην συρρήκνωση της, έρω της ενιαίας αγοράς. Έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες. Οι περισσότερες αναφέρονται στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για όλα τα μέσα μεταφοράς και ζήτησα από την Επίτροπη να συντάξει μία έκθεση σε σχέση με τις δημόσιες μεταφορές σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης ζήτησα να διασφαλίσουμε τις σωστές κοινωνικές συνθήκες και κοινωνική ισότητα ως προς την χρήση των μεταφορών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης υπέβαλα μία τροπολογία που αναφέρεται στον ταχυδρομικό τομέα. Γιατί εάν λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να απελευθερώσουμε τις ταχυδρομικές μεταφορές και έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις κοινωνικές συνθήκες ισομέρειας. Εδώ αναφέρομαι και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και ζήτησα μέσω μιας τροπολογίας από την Επιτροπή να μας κάνει μια γενική παρουσίαση για τις εταιρίες low cost, δηλαδή κατά πόσο πλήττουν άλλες μεταφορές. ιδιαίτερα όταν λειτουργούν από ορισμένα αεροδρόμια και ζήτησα να προβεί σε έναν υπολογισμό για τους επίναυλους και την μεταφορά των αποσκευών των επιβατών. Αυτό αφορά τις εταιρείες low cost. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς την πραγματική χρήση των χρονοθυρίδων και αυτό αφορά τις εναέριες μεταφορές βεβαίως αποκλειστικά. Παράλληλα, ένα τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η αίτηση προς την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα πρότασης ορισμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τις λιμενικές αρχές να εξασφαλίσουν τις θαλάσσιες μεταφορές. Διότι δυστυχώς οι θαλάσσιες μεταφορές δεν έχουν ενισχυθεί όπως θα έπρεπε τον τελευταίο καιρό. Ο κύριος Τέρξ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη συνεργασία. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ε, διατρανωθεί η θέλησή μας, διότι θα πρέπει να έχουμε έναν εξισορροπημένο τρόπο μεταφορών, εξισορροπημένο ως προς τα διάφορα μέσα για την ανάπτυξη της οικονομίας. Συμφωνώ με την πρόταση συμβασμού υπαριθμών Α ως προς τις προτεραιότητες. Συμφωνώ λοιπόν με την τροπολογία συμβιβασμού υπαριθμών 1. Ο συνάδελφος Μούλντε προέβαλε τις τροπολογίες 15, 16, 17, 18, 26 και 28 για τις 15 και 16 Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εξορρόπηση μεταξύ ε, φόρων και εισφορών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι 15 και οι 16 είναι, οι τροπολογίες 15 και 16 είναι σωστές. Δεν ξέρουμε πώς δαπανώνται όμως αυτά τα χρήματα. Ως προς τα δικαιώματα των ε, επιβατών, δεν ξέρω κατά πόσο εμπίπτουν στην πολιτική ανταγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να πούμε ότι όλα τα μέσα μεταφοράς, μάλλον ε, ναι, όλοι οι τρόποι μεταφοράς, το διατροπικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να οδηγεί σε δικαιώματα, δηλαδή μία ώρα χρήσης είναι διαφορετική, ανάλογα με το ποιο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει τις τροπολογίες 21 και 22. Λέμε να είναι δίκαιοι, αλλά όχι ίση, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα εδώ ως προς τις αντισταθμίσεις. Ως προς την ε, τροπολογία 19, ε, γίνεται λόγος για equal, ίση αντιστάθμιση δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει ε, αντιστοιχεία, αντιστοίχηση με το Ολλανδικό κείμενο. Ως προς τις 27 ε, και 28 το καμποτάζ, πιστεύω ότι πολλές φορές ε, υπάρχουν εμπόδια για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ως προς το καμποτάζ. Επίσης, ως προς τις επιδοτήσεις λιμένων, τις επιδοτήσεις τις περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Θα πρέπει να προωθηθούν. Γιατί περιμένει η Κομισιόν. Ως προς τις, ε, τα ταχυδρομικά συστήματα, ε, συμφωνώ με την κυρία Τσικάου ως προς το κείμενο, δηλαδή να λάβουμε το κείμενο από την οδηγία για τις ταχυδρομικές μεταφορές, όχι μόνο τις κρατικές επιδοτήσεις, αλλά να έχουμε και μία υψηλή κοινωνική προστασία. Αυτά λέει η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Για την τροπολογία συμβασμού Β συμφωνούμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την εργασία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι, σιδρο, οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν μέτρο σύγκρισης. Δεν αποτελούν το μέτρο. Δεν είναι ε, σωστός ο όρος σύγκρισης. Εμείς προσπαθήσαμε να εξορπίσουμε αυτή την ε, ε, έκθεση με αυτές τις τροπολογίες. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω, ακούγοντας τη συζήτηση, ότι το καμποτάζ είναι η πιο ε, το πιο διακριτικό τμήμα ε, κάθε συνθήκης προσχώρησης. Το καμποτάζ, οι κανόνες του καμποτάζ ε, προκαλούν διακρίσεις και ε, νομίζω ότι είναι αντίθετες προς μία από τις τέσσερις ελευθερίες που είναι στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καμποτάζ είναι ένα βασικό θέμα. Αν υπάρχουν εμπόδια στο σύστημα του καμποτάζ, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για ελεύθερο ανταγωνισμό, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για αποτελεσματικότητα στις μεταφορές εμπορευμάτων και αγαθών. Αν παραδείγματος χάρη ένα φορτηγό τσέχικο ε, ταξιδεύει προς την Ισπανία, ε, θα πρέπει να γυρίσει άδειο ε, πίσω στην χώρα του. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Και μιλώντας για κοινωνική προστασία, για ίσες όρους, ίσες συνθήκες, έχουμε κάνει πολλά, αλλά όχι όλα. Σχετικά με τα πλοία, τα πλοία είναι ένα περιβαλλοντικό μέσο μεταφοράς, κυρίως εσωτερικές υπηρετικές ε, μεταφορές ε, στη Βόρεια Γαλλία, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε ε, το Δούναβι, ο οποίος είναι ο μακρύτερος ποταμός της Ευρώπης. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε μέσα στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα, αλλά είμαι ευγνώμων που αναφέρονται τα κοινωνικά θέματα για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι σημαντικό, διότι προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε τις μεταφορές θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, τις κοινωνικές συνθήκες, την κοινωνική προστασία και τις ευκαιρίες για θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι ε, το συμβιβασμός θα είναι καλός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Κρέμερ για την εισήγηση και δεν μπορώ παρά να πω ότι στην ομάδα μου δεν θα είναι εύκολο να βρούμε μια λύση για την έκθεσή σας, αλλά θα κάνουμε το παν. Τώρα σε σχέση με ορισμένα ειδικά σημεία. Ο κύριος Στέρκ ανέβηρε ήδη ορισμένα σημεία σχετικά με την επιθυμία σας να εισαγάγετε αποζημιώσεις για τις σας στους σιδηροδρόμους. Βεβαίως, ο χρόνος είναι χρήμα και πρέπει να υπάρξει αποζημίωση για την απώλειο χρόνο, αλλά αυτό το μεταφορικό μέσο είναι διαφορετικό και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη το τι πληρώνουμε για το σιδηρόδρομο και για το τι πληρώνουν οι επιβάτες για τις δρομικές μεταφορές. Νομίζω ότι οι αποζημιώσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο μέσο αυτό. Μην προχωρήσετε τόσο πολύ και να ακούστε άλλους συναδέλφους που ζήτησαν μια πιο, πιο μετριοπαθή προσέγγιση σχετικά με το άρθρο 7 πολλοί θέλανε να γράψουν κάτι σε σχέση με το θέμα αυτό. Σας υποστηρίζω εγώ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες αν μπορεί η Επιτροπή να έχει μια τέτοια έκθεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υποστηρίζω την τροπολογία 30 σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να υπάρχει έκθεση για τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εργάζονται μόνο για τρία χρόνια, δηλαδή που είναι νέες εταιρείες. Θα πρέπει να δούμε τις εταιρείες χαμηλού κόστους που έχουν συμβάσεις δεκαετίας και άνω. Σχετικά με το dumping, χαίρομαι που ζητείτε μια πλήρη απελευθέρωση στον τομέα αυτών. Ε, είμαι μαζί σας και πιστεύω ότι και η ομάδα ALDE είναι μαζί μας σχετικά με το θέμα αυτό, διότι το κοινωνικό dumping είναι πάρα πολύ άδικο ε, και αξίζει να έχουμε μια διεξοδική συζήτηση. Αλλά η παρούσα κατάσταση, η κρίση στα νέα ε, κράτη-μέλη, το επίπεδο των μισθών έχει πέσει πολύ και είναι χαμηλότερο από ό,τι πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άλλα κράτη-μέλη ε, κλείνουν αυτόν τον τομέα μεταφορών και έτσι ε, υπάρχει περισσότερο dumping και δεν έχουμε κοινωνικές εγγυήσεις στα νέα κράτη-μέλη, διότι υπάρχει μεγάλο άνοιγμα ε, στις μισθούς, στις αμοιβέ ανάμεσα στα νέα κράτη-μέλη και στα παλιά. Χρειαζόμαστε τότε έναν φόρο επί του κεφαλαίου για την απόκτηση αγροτικής γης, παραδείγματος χάρη Όλα αυτά εξαρτώνται από την ικανότητα να ε, μπορεί κανείς να έχει πιστώσεις, ε, δάνεια και τα επιτόκια διαφέρουν ανάμεσα στις παλιές χώρες και στις νέες χώρες. Όλα αυτά επανέρχονται στο κοινωνικό dumping. Νομίζω ότι τότε θα έχουμε μια πλήρη κατατεμαχισμό ε, της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ευχαριστώ κύριε Ρίκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μάικλ Κράμερ, ο οποίο με στεναρότητα ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σα πάνω σε τρει τροπολογίες 36 και 37 που καταθέσαμε, διότι νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε τις έμεσες επιπτώσεις λόγω των κανόνων πιστοποίησης, λόγω των κανόνων ασφαλείας που οδηγούν σε διακρίσεις και θα πρέπει να επισύρω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στα προβλήματα αυτά στον τομέα των σιδηροδρόμων. Τα δεύτερη και τελευταία παρατηρήσή μου δεν θα σας εκπλήξει, αναφέρεται στην τροπολογία 18 του κ. Κρέμερ. Θα μπορούσα να πω ότι λυπήθηκα ως Γάλλος διότι μας αναφέρει ονομαστικά αλλά δεν είναι αυτή η παρατήρηση που θέλω να κάνω. Θα ήθελα να κάνω πολλές παρατηρήσεις ως προς την ουσία του πράγματος. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι υπενθυμίζω ότι η έκθεση αναφέρεται στο 2009 και ο φόρος που αναφέρεται στην τροπολογία 18 δημιουργήθηκε το 2010. Ήδη υπάρχει λοιπόν ένα μικροχρονικό λειτουργικό πρόβλημα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν ε, ανακρίβειες αρκετά σημαντικές στην τροπολογία αυτήν. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον φόρο ε, για τα δίκτυα και την κατάργηση του trade tax, ε, μέτρο που είναι ξεχωριστό χρονικά και ως προς την ουσία. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην διαγραφή του ενός και την εισαγωγή του άλλου φόρου. Επίσης, ο φόρος δεν αναφέρεται ε, μόνο στα μέσα μεταφοράς, αλλά για το σύνολο των δικτύων, ε, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ε, και είναι δύσκολο να τοποθετηθεί εδώ σε αυτήν την τροπολογία. Τρίτη παρατήρηση ως προς την ουσία είναι ότι αυτό το είδος του φόρου υπάρχει σήμερα σε πάρα πολλές χώρες και συνεπώς δεν είναι κάτι το ειδικό όπως θα νόμιζε κανείς από την τροπολογία. Τέταρτη παρατήρηση είναι ότι έχει επιληφθεί του θέματος η Επιτροπή για το θέμα αυτό και το φόρο και δεν, δεν θα επισύρουμε την προσοχή της εφόσον τα εξετάζει αυτά. Την, για να δούμε αν το κείμενο αυτό είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους η ομάδα μου θα ήθελε να καταθέσει μια προφορική τροπολογία για την τροπολογία 18 που μπορώ να σας διαβάσω στα αγγλικά που είναι μια τροπολογία στη θέση αυτής που περίπου λέει τα ίδια πράγματα αλλά με το τρόπο που καλύπτει τις διάφορες παρατηρήσεις που έκανα για την μορφή και την ουσία. Ζητεί από την Επιτροπή να βεβαιωθεί ότι η φορολόγηση εθνική δεν αποτελεί εργαλείο διακρίσεων εναντίον των ξένων εταιριών στον τομέα των μεταφορών. Αυτό προτείνουμε. Ευχαριστώ. Ελπίζω στη γραμματεία να κατέγραψε την τροπολογία σας. Ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι άλλοι ομιλητές, συγχαίρω τον κύριο Κρέιμερ που έκανε πολλή δουλειά, επιθυμητή και φιλόδοξη. Αν και οι στόχοι θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν, κυρίως θα μιλάμε για την ισχύ των ίδιων κανόνων σε όλο το σύνολο του μεταφορικού τομέα. Συμφωνώ με τα σχόλια του κυρίου Στέρκ και ενός ή δύο άλλων μελών σε ό,τι αφορά την τροπολογία 21. 25% αποζημίωση καθυστέρηση μια ώρα, 5% για καθυστέρηση πάνω από δύο ώρε σύμφωνα με την ισχύ νομοθεσία στο μέσο των δρομικών μεταφορών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι για το θέμα της αποζημίωσης, αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί Μιλάμε για σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες για τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να ισχύσει επίσης μία αποζημίωση. Οι σιδηρόδρομοι, ε, ναι, έχουμε τους σιδηροδρόμους αφενός, αλλά υπάρχουν και άλλες μεταφορικές υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θέλουμε να ανοίξουμε ε, ε, την, τη δημόσια, την υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος και σε ό,τι αφορά τα ταχυδρομεία. σε ό,τι αφορά τις κρατικές εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, αν φτάσουν στην αγορά, στην αγορά ε, άλλες εταιρείες, θα υπάρξουν σοβαρές επικαλύψεις. Γι' αυτό με ικανοποιεί αυτή η τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, περίμενα να τελειώσει η διερμηνία. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέιμερ για τη δουλειά του και να αναφερθώ σε δύο ή τρία σημεία. Πρώτον, την αρχή της αμοιβαιότητας που αναφέρεται στην τροπολογία 35. Καταρχήν συμφωνώ με αυτή την αρχή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η αρχή της αμοιβαιότητας θα είναι κάτι το μεταβατικό και όχι κάτι το μόνιμο τροπολογία, σχετικά με την τροπολογία όσοι έχει τώρα, υποστηρίξαμε το αρχικό κείμενο, αλλά θα θέλαμε αυτό να εκφράζει σαφέστερα αυτό που ελέγχθη στην Επιτροπή. Είτε θα δεχθούμε εταιρείε που συμμετέχουν στι αγορέ άλλων κρατών μελών εκτός των δικών τους δεν είναι σαφής η διατύπωση εδώ. και υπάρχει πολλές αγορές είναι κλειστές και δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής εταιριών από άλλες χώρες. Σε πολλές επίσης χώρες υπάρχουν ορισμένα μονοπόλια τα οποία δεν έχουν ακόμα καταργηθεί με αποτέλεσμα άλλες εταιρείες να αποκλείονται από αυτές τις αγορές. Θα χρειαστεί να βρούμε μια διατύπωση η οποία να ανταποκρίνεται σε αυτό που πρεσβεύουμε σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Και για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες προφανώς όλα θα εξαρτηθούν από τις ε, αρμοδιότητες. Υπάρχουν προβλήματα για την ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Τώρα για το φόρο στη Γαλλία. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούμαστε να δούμε αυτό το θέμα, να συζητήσουμε αυτό το θέμα γραπτός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο νόμος τον οποίο αναφέρεστε δεν είναι το πρόβλημα από την άποψή μου. Υπάρχουν άλλοι νόμοι που εξακολουθούν να ισχύουν στη Γαλλία και οι οποίοι διονίζουν μονοπωλιακές καταστάσεις σε ορισμένους τομείς. Και θα πρέπει να δούμε, όταν καθιερώθηκε η Ευρωβινιέτ, ορισμένες χώρες είπαν ότι όλοι πρέπει να έχουμε ευρωβινιέτ και θα αποδίδουμε τα χρήματα στους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν κατά την άποψή μου να υποστηρίξουμε την προφορική τροπολογία είναι σημαντικό να αναλύσουμε όλους τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε στρέβλωση, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Αυτά είχα να πω εξ ονόματος της ομάδας και ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπαμε, χαιρετίδη, μας ικανοποιεί η εργασία του κυρίου Κρέιμερ και λάβαμε γνώση των συστάσεων. Τώρα, γιατί θα θέλαμε να κάνουμε την εξή δήλωση. Η Επιτροπή είναι υπέρ της προοδευτικής του προοδευτικού ανοίγματο και τη απελευθέρωση τη αγορά των σιδηροδρόμων. Όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη ενό ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξετάζει τις επιπτώσεις του και τη σημασία του κανονισμού 1370. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβεί σε μία αξιολόγηση των ωφελών και των εξόδων για, τη, για όλους τους τομείς των μεταφορών το 2011 ώστε να προωθήσει την περαιτέρω, το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών. Θα ε, καλύψει αυτό το άνοιγμα τη ε, μεταφορά ιδιωτών με την παροχή και την εξασφάλιση των κατάλληλων εχέγγυων. Κατά γενικό κανόνα, ο κανονισμός 1370 του 2007 επιτρέπει την ε, κατακύρωση συμβάσεων χωρίς ε, δημόσιο διαγωνισμό. Αυτός ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη συμμετοχή των σιδηροδρομικών εταιριών σε διαγωνισμούς Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προτινόμενες τροπολογίες, θέλουμε να προσθέσουμε ορισμένες περαιτέρω διευκρινήσεις. Τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται και εγκρίνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφιστά την προσοχή των μελών στο scoreboard που δημοσιεύει δύο φορές το χρόνο, άνοιξη και φθινόπορο, και αναφέρομαι στις τροπολογίες 5 και 9. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την τροπολογία 9, οι κατευθυντήριε γραμμές για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις ισχύουν, εφαρμόζονται επίσης και στον κανόνα των μεταφορών. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την παράγραφο την τροπολογία, συγγνώμη, διορθώνει μιλήτρια 40, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καθιερώσει κατευθυντήριε γραμμέ για τι ενισχύσει στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Τροπολογίε τροπολογίες 30 και 31 που αναφέρονται στις περιπτώσεις τοπικών μεταφορέων. εξ ορισμού του, αυτού του είδους οι ενισχύσεις δυνητικά θα μπορούσαν να αποδειχθούν ασυμβίβαστης και γι' αυτό τα κράτη-μέλη δεν ε, ε, εμφανίζουν με απόλυτη διαφάνεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτού του είδους ενισχύσεις. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 41 και 43, ε, κατευθυντήρες γραμμές για τις ενισχύσεις στα λιμάνια. Θα ξεκινήσει μια μελέτη του επόμενου τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, εξετάσει την κατάσταση και να αποφασίσει τι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εφαρμοστούν. Θέλετε να επανέλθετε. Εντάχει. Νομίζω ότι ξέχασα το θέμα της αμοιβαιότητας. Θα ήθελα να πω έμπρακτα μόνο αυτό που θεσπίστηκε στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Αυτό ήθελα να εκφράσω. Εν πάση περιπτώσει θα διορθώσω τα δεδομένα αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση γιατί εγώ είχα δώσει μεγάλη μάχη έτσι ώστε οι γαλλικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να δράσουν στη γερμανική αγορά, να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτός ήταν ε, ο αρχικός μου σκοπός, απότερος σκοπός. Τη στιγμή που στη Γερμανία υπάρχει ε, ρύθμιση του τομέα των σίδεροδρόμων μέσα στα πλαίσια του, της Deutsche Bahn μπορέσαμε να αλλάξουμε τον κανονισμό το υπόβαθρο. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να μην αναφέρουμε τη λέξη Γαλλία, αλλά ας ε, μιλήσουμε για τους φόρους όπως θα ισχύσουν. Για την τροπολογία 10... Mein Vorschlag besser. Aber... Για την τροπολογία 10 η πρότασή μου είναι η καλύτερη νομίζω. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή σε σχέση δηλαδή με τις πλωτές οδούς και τους ε, σιδηροδρόμους καθώς και τις πολιτικές ε, τιμολόγησης. Δεν θα ήθελα για τις καθυστερήσεις να καταβάλουν μεγάλο αντίτιμο οι επιχειρήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις εις βάρος του επιβάτη. Στο Βερολίνο αυτές τις αντισταθμίσεις ε, ορίσαμε σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και ιδιαίτερα μεγάλων καθυστερήσεων. Έχουν οριστεί σε τοπικό επίπεδο τη στιγμή δηλαδή που οι επιβάτες έχουν, αντιμετωπίζουν μεγάλη καθυστέρηση να μπορούν να πάρουν ένα ταξί ας πούμε και να καταβληθεί το αντίτιμο σε αυτή την περίπτωση. Άρα η βασική ιδέα είναι να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να μην ε, επιλέγουν το κέρδος αποκλειστικά, αλλά να προβάλλουν και υπηρεσίες ακριβίας και να μην ζημιώνουν, εν πάση περιπτώσει, τον επιβάτη. Ως προς τις ε, ταχυδρομικές ε, υπηρεσίες, μπορώ να σας πω στη Γερμανία ότι ο, ο γιος μου εργάστηκε στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας, αυτή την υπηρεσία και αυτά που είδε σε μία τέτοια ΜΜΕ ήταν ανατριχιαστικά. Θα θέλαμε να δούμε πού υπάρχει dumping και όπου υπάρχει να διαγραφεί να απομακρυνθεί βεβαίως. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους σιδηροδρόμους για να φτάσουμε στους οικολογικούς μας στόχους. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής οι οδικές μεταφορές υποστηρίζονται ιδιαίτερα εις βάρος των σιδηροδραμικών ως προς την μετάβαση, το πέρασμα των συνόρων, έλαβα συγκεκριμένες επιστολές όπου αναφέρεται ότι στην περίπτωση έγκρισης δεν θα υπάρχουν διακρατικές μεταφορές γιατί οι φόροι στα σύνορα είναι πολύ υψηλοί και θα αποθαρρύνουν τις μεταβάσεις αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο φορολόγησης. Ε, χαίρομαι ε, που προβάλλει στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ιδιαίτερα, αύριο θα ψηφίσουμε στις 30 Νοεμβρίου στη συνέχεια και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Το επόμενο θέμα ελπίζω να το δούμε γρήγορα, διότι αναμένουμε και την Επίτροπο την κυρία Δαμανάκη να συζητήσουμε. Είναι η δική μου έκθεση για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού θα ήθελα να κάνω ορισμένα γενικά σχόλια. Ξέρετε ότι είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις και αναγνωρίζω ότι θα... Ε, νομίζω ότι θα υπάρξει ομοφωνία, υπάρχουν όμως, ανακύπτουν όμως ορισμένα ζητήματα. Θεωρώ θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για να έχουμε ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού μέσα στα πλαίσια της συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης στα κράτη-μέλη. Όμως, ως προς τις κατεξουσιοδότηση ε, εξουσίες που προβλέπονται, κατεξουσιοδότηση υποχρώσεις, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ορίσουμε τις κατεξιοδότηση πράξης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την τακτική νομοθετική διαδικασία και γι' αυτό προτείνω μια σειρά τροπολογιών για τον περιορισμό των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων αυτών. Επίσης, ε, δεν ε, Είμαι υπέρ των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες για να ξέρουμε πώς έχει η βιομηχανία τουρισμού στο σύνολό της και πώς συγκρίνεται με άλλους τομείς βιομηχανίας καθώς και οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση. Γι' αυτό θα πρέπει να εισαχθεί μια διάταξη έτσι ώστε τα κράτη να διενεργήσουν πιλωτικές έρευνες σε σχέση με τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό και εάν χρειαζόμαστε εναρμονισμένους πίνακες, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Ως προς τα, τις τροπολογίες των μελών θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες όπως προβάλλουν οι σοσιαλιστές οι πράσινοι και οι, ως προς τις ε, τροπολογίες της τροπολογίας του κ. Φιντάνσε. Όμως η τροπολογία 13 σε σχέση με τις στατιστικές για το catering, για υπηρεσίες catering, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί, αλλά επειδή μίλησα με την Προεδρία, ε, δεν είναι σαφές τι εννοούν σε σχέση με ε, αυτή την ιδέα για τον τομέα της εστίασης και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μία ξεχωριστή έκθεση ή μελέτη για το τομέα της εστίασης όπως ορίζει η τροπολογία Φιντάντσα. Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία Φιντάντσα και άλλων, αν και θα ήθελα να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας πει τι μπορεί να εφαρμοστεί εδώ. Εν πάση περιπτώσει, η Προεδρία θεωρεί ότι το Συμβούλιο δεν θα δεχόταν αυτό το διαχωρισμό στατιστικών στοιχείων. Επίσης, αντιτίθεμε στην τροπολογία Κόσα, διότι αυτές οι τροπολογίες δεν λαμβάνουν υπόψη τον ημερήσιο τουρισμό. Και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ε, μην λάβει υπόψη το μονοήμερο τουρισμό. Υπάρχουν όμως άλλες τροπολογίες από άλλες ομάδες και μεμονωμένα μέλη που μπορώ να υποστηρίξω. Άρα το μόνο πρόβλημα για μένα είναι η τροπολογία 32 του κυρίου Φιντάντσα σε σχέση με τον τομέα της εστίασης και τα ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία για τον τομέα της εστίασης. Ο κύριος Φιντάντσα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή εργασία και για τις βασικές αρχές τις οποίες αναφερθήκατε και η ομάδα μας συμφωνεί ως προς τις κατεξιοδότηση πράξης συμφωνούμε και εμείς ότι αυτές είναι οι βασικότερες αλλαγές στην τακτική διαδικασία. Γι' αυτό θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες σας. Επίσης θα υποστηρίξουμε και τις τροπολογίες που σχετίζονται με τις μονοήμερες εκδρομές. Θα ήθελα να σας πω ότι 21, 23 και 24 τον, του συναδέλφου Κόζα θα αποσυρθούν. Δέχτηκε ο συναδέλφος να τηρηθεί ε, αυτή η αρχή, να λάβουμε υπόψη δηλαδή τις μονοήμερες εκδρομές και εγώ υπέβαλα και την τροπολογία 22 για να ορίσουμε καλύτερα τις ημερήσιες επισκέψεις. Και θα ήθελα να σας πω, συνάδελφοι, ότι υπάρχει και μία προφορική τροπολογία που υποστηρίζει την 22 τη διαβίβασα στη γραμματεία και είναι μία προσαρμογή της ορολογίας καθαρά σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιούμε σε άλλα σημεία του κειμένου. Ελπίζω να δεχτείτε αυτή την προφορική, η οποία απλώς διορθώνει την σύνταξη. Ως προς τις 8 και 25, εμείς θα υποστηρίξουμε την 8 του εισηγητή, άρα 25 θα καταπέσει και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με την 26 του συναδέλφου Κόζα, όπου ορίζουμε μία ημερομηνία θέσεως ισχύ, δηλαδή όταν συλλεγούν οι πληροφορίες και μετά από συμφωνία με τον κύριο Κόζα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποβάλουμε άλλη μία προφορική ως ΕΛΚ για να ορίσουμε μία ημερομηνία για την αρχή συλλογής δεδομένων δηλαδή σε περίπτωση αναθεώρησης του κανονισμού. Δεν μιλάμε για την πρώτη εφαρμογή βεβαίως, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2012. Αλλά σε περίπτωση αναθεώρησης, αν η νομοθετική διαδικασία δεν λήξει στις 30 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε κερδίζουμε ένα χρόνο. Ε, δηλαδή το μεταφέρουμε ένα χρόνο μετά έτσι ώστε οι ΜΜΕ που συμμετέχουν στον τουρισμό να είναι σε θέση να συλλέξουν πληροφορίες. Θεωρούμε ότι αυτή η διατύπωση που είναι διαφορετική από την αρχική του κυρίου ε, Κόζα που μιλούσε για τις 30 ε, Ιουνίου του έτους έναρξης ισχύω, μας οδηγεί σε ένα κέρδος τριών μηνών έτσι ώστε θα είναι δυνατόν, να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός. Εμείς θα υποστηρίξουμε, γιατί στην 27 βλέπω ένα πλήν του συνάδελφου Κόζα, εμείς όμως θα θέλαμε να υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία που αποσκοπεί στην απλούστευση των κατηγοριών και των ε, τρόπων και λόγων ταξιδίου όταν μιλάμε για προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς. Ως προς, ε, την τροπολογία 32 για τα εστιατόρια, την υπέβαλα μόνο για να υπάρχει συνοχή του κειμένου, διότι γνωρίζουμε οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν γνωρίζουν ότι το θέμα αυτό εισήχθη ήδη στο παράρτημα που αφορά τις ημερήσιες επισκέψεις. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη αξία στις ε, στατιστικές αναλύσεις των ε, ημερησίων επισκέψεων. Γι' αυτό χρειάζεται αυτός ο δείκτης και για, τις, ε, και για τη διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν είναι θέμα ζωής ή θανάτου βεβαίως. Νομίζω όμως ότι για λόγους συνοχής και επειδή το θέμα είναι σημαντικό, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό τον επιμερισμό και για τον, ε, και για τον τυρισμό και σε σχέση με τις επισκέψεις μικρής ή μακράς διάρκειας θα θέλαμε να την κρατήσουμε αυτή την τροπολογία. Και αν υπάρχουν και άλλες υποδείξεις, ευχαριστώ να τις ακούσουμε. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος κάποιου άλλου που δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Θα είμαι ε, σύντομη συμφωνούμε με τα περισσότερα σημεία τα οποία τονίσατε. Υπάρχουν και μερικά με τα οποία δεν συμφωνούμε. Τροπολογία 27 νομίζω ότι είναι ευστοχή αυτή η μείωση και για το λόγο αυτό θα δεχθούμε την 27 για την 31 και εδώ επίσης συμφωνούμε διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και επίσης συμφωνούμε με τα όσα είπε το ΕΛΚΑ για όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τα παρουσιάσατε πάρα πολύ καλά, τα ρυθμίσατε πάρα πολύ καλά και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας σχετικά με τα σημεία αυτά. Κυρία Ντιουράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εισηγητά. Ευχαριστώ για την καλή σας εισήγηση. Θα ήθελα ε, για μερικές τροπολογίες να, να υπενθυμίσω για την τροπολογία 25 που καταθέσαμε και για την οποία ζητούμε όχι μόνο το περιβάλλον, ο αντίκτυπος για το περιβάλλον να ληφθεί υπόψη, αλλά και ο αντίκτυπος ε, πάνω στην ε, κλιματική αλλαγή, δηλαδή οι εκπομπές. Δεν καταλαβαίνω, στις ψηφοφορίες ζητάτε να ψηφίσουμε πρώτα την 8 και μετά την 25, αλλά νομίζω ότι η 25 προχωράει πολύ περισσότερο από την 8. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και μετά, αν δεν ψηφιστεί, ε, να περάσουμε στην 8, διότι νομίζω ότι η 25 είναι ακριβέστερη, ζητάει να μετρηθούν οι επιπτώσεις πάνω στην κλιματική αλλαγή ε, και να δούμε την εφαρμογή διάφορων οικοσημάτων, ε, οικοσημάνσεων Γι' αυτό ζητώ από τους συναδέλφους να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία πάνω στο γεγονός βεβαίως ότι η μέτρηση πάνω στο περιβάλλον τροπολογία του κυρίου Σίμψον είναι σημαντική, αλλά εφόσον αυτό είναι γενικό, ζητούμε στην τροπολογία 25 τις επιπτώσεις ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά για τις μεταφορές. Είναι ε, σημαντικό, οι άνθρωποι πήγανε με αεροπλάνο, με τρένο, με αυτοκίνητο, στον τουριστικό προορισμό, με τα πόδια ή με το ποδήλατο είναι σημαντικό να το ξέρει κανείς ως πληροφορία. Δεύτερο πράγμα, η τροπολογία που αναφέρεται ε, στην, στο παράρτημα 2.1.1 η χρησιμοποίηση των ποδηλάτων όχι μόνο για να πάει να διακοπές διότι υπάρχουν πολύ λίγοι που πάνε διακοπές με ποδήλατο αλλά υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί φεύγει κανείς με το αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο ή πάει κανείς ε, με το αυτοκίνητο και μετά νοικιάζει κανείς ε, ε, ένα ποδήλατο είναι σημαντικό ε, που και σε ποια περιοχή χωρίς να ασκήσουμε πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μεγάλες οι επενδύσεις για τις μικρομεσαίες, θα πρέπει να υποστηρίξουμε πολιτικές διαρρύθμισης, ανάπλασης διαφόρων χώρων για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Και αυτό είναι καλό όχι μόνο για τα άτομα αυτά, αλλά και για τις οικογένειες. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε αυτές τις τροπολογίες και ελπίζω ότι θα έχουμε την υποστήριξη σας. Ο κύριος Ντιμούντα για την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την υποστήριξη για την, τον κανονισμό γενικά και για την εισήγηση και για την δεύτερη σειρά τροπολογιών που λάβαμε πρόσφατα σχετικά με το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Νομίζω ότι τα όργανα βρίσκονται στην ίδια γραμμή περίπου. Συμφωνούμε με την γραμμή που ακολουθήθηκε και όσον αφορά τις τροπολογίες 2, 3, 5, 6, 7, 10, δεν, 16, ε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για να καταλήξουμε σε συμφωνία. σχετικά με τα πιο τεχνικά πράγματα. Ακούμε με ευχαρίστηση ότι οι τροπολογίες 21, νομίζω 23 και 25 πιθανόν δεν θα υποστηριχθούν ε, διότι στην εισήγηση είδαμε ε, τι έχει εισαχθεί και με τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να περιβάλλουμε, να περιλάβουμε κάτι για τις μονοήμερες υποσκέψεις. Τα κράτη-μέλη επίσης φαίνεται ότι συμφωνούν σχετικά με την συμπερίληψη των μονοήμερων επισκέψεων. Σχετικά με την τροπολογία νομίζω 22 για τον ορισμό για τις επισκέψεις τις μονοήμερες, με έκλειψη είδαμε ότι προσθέθηκε μια ανασορισμός διαμέσου μιας τροπολογίας, διότι στο άρθρο 4-5 βλέπουμε ποιο είναι το πεδίο αυτό, το πεδίο εφαρμογής για τις μονοήμερες επισκέψεις. Λέμε ότι πρόκειται για επισκέψεις, για ταξίδια εκτός του τόπου κατοικίας που διαρκούν μια μέρα θα πρέπει βεβαίως αυτές οι επισκέψεις να αρχίζουν ε, από τον, ε, τον τόπο κατοικίας. Τροπολογία 22. Δεν είμαστε πεπισμένοι για την χρησιμότητα του ορισμού στο άρθρο 2. Καλύτερα να έχουμε ένα πεδίο στο άρθρο 4 παράγραφο 5. Επίσης, το στοιχείο της α, ανάπαυλας, ε, της ψυχαγωγίας, της αναψυχής. Ε, δεν νομίζω ότι ε, φιλοδοξία των στατιστικών τουρισμού είναι να μετρούν αυτές τις μονοήμερες εκδρομές για να μείνει κανείς σε μια πισίνα ή δεν ξέρω τι. Άλλο είναι οι τουριστικές μονοήμερες επισκέψεις. σχετικά με τις τροπολογίες 18 και 25 για την οικολογική σημασία του τουρισμού. Νομίζω ότι σε σχέση με την τροπολογία 18 που αναφέρεται στο εκτιμώντας 6 υπάρχει ε, μία, ένα πρόβλημα με την διατύπωση οικολογικής οικολογική σημασία με βάση το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό. Αυτό το αποδεκτό πλαίσιο αναφέρεται μόνο στον οικονομικό αντίκτυπο του τουρισμού ενώ ε, το πλαίσιο αυτό για τους δορυφορικούς λογαριασμούς δεν είναι το κατάλληλο για να μετρηθεί η οικολογική σημασία. Υπάρχουν μερικές ασκήσεις στην Δανία, στη Σουηδία που έχουν κάνει προκαταρκτική εργασία για να συνδέσουν με τους, ε, τους τουριστικούς λογαριασμούς, με δορυφορικούς λογαριασμούς ε, οικολογικούς και για τον τουρισμό. Νομίζω ότι υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με τα αυτά που αναφέρονται στον, στο εκτιμώντας 6 και στην τρέχουσα πρακτική, στην αιτιολογική σκέψη 6. Έχουμε και την τροπολογία 25. Επίσης εδώ αυτό δεν ε, σχετίζεται με τους ε, δορυφορικούς λογαριασμούς του τουρισμού. Είναι κάτι που είναι αποδεκτό από τον, ε, τον το Οργανισμό Τουρισμού, αλλά για το Eurostat δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούμε να περιλάβουμε οικολογικές απόψεις. Η ιδέα του να έχουμε πιλωτικές μελέτες για να έχουμε μια καλύτερη άποψη σχετικά με τον αντίκτυπο του τουρισμού πάνω ε, στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο. Μια προειδοποίηση θα ήταν ότι θα πρέπει ίσως να μην απομακρυνθούμε πολύ από το πεδίο του τουρισμού, διότι είναι ένας, ε, μια, ένας κανονισμός για τις στατιστικές ε, περί τουρισμού. Δεν πρέπει να ε, περιλάβουμε την ενέργεια, το περιβάλλον, τόσο πολύ τις μεταφορές πρόκειται για τον τουρισμό. Το σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η μέτρηση του τουρισμού των στοιχείων του τουρισμού και των δευτερογενών επιπτώσεων βεβαίως σχετικά. Τώρα περνάω. Ε, πήγα από την 25 στη 18 διότι σχετίζονται η τροπολογία 19 ε, στοιχεία για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην τρέχουσα ε, πρόταση στο 1β του παραρτήματος υπάρχει υπάρχουν οι κοινωνικοί λόγοι για τη μη συμμετοχή στον τουρισμό. Υπάρχουν μερικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό σχετικά με τα στοιχεία για ειδικέ ομάδες, υπερήλικες, άτομα με ειδικέ ανάγκες, νέα άτομα. Ίσως υπάρχει πρόβλημα από τεχνικής απόψεως για το πώς είναι οργανωμένες οι υπηρεσίες. Υπάρχουν περιορισμένες υπηρεσίες για 5.000, 10.000 και έχουμε δειγματοληπτικές έρευνες οι οποίες δεν είναι επαρκείς για την παραγωγή καταλήλων στατιστικών για διάφορες ομάδες. Και είναι δύσκολο να περιληφθούν σε αυτήν την έρευνα. Μια λύση θα ήταν να διευρύνουμε την έρευνα και να περιλάβουμε περισσότερα άτομα, αλλά αυτό θα είχε επιπτώσεις πάνω στον προϋπολογισμό και στο κόστος που είναι απαράδεκτο. Είναι κάτι βεβαίως που θα πρέπει να το εξετάσει το Συμβούλιο. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στο τμήμα 1β. Υπάρχουν επίση άλλες στατιστικές, στατιστικές για το, το, το βιωτικό επίπεδο, τα εισοδήματα αν ε, μια οικογένεια μπορεί να έχει διακοπές μία φορά το χρόνο, μία εβδομάδα. Ε, για την τροπολογία 19 έχουμε προβλήματα συλλογής ε, στοιχείων, δυνατότητας να έχουμε αξιόπιστες στατιστικές για μικρές σχετικά ομάδες της κοινωνίας, διότι τα δείγματα ίσως δεν είναι αρκετά επαρκή. Σχετικά με την τροπολογία 20, κύριε Ντιμόντε, Έχω μια επίτροπο έξω που περιμένει ε, και... Ναι, θα σας ζητούσα λοιπόν να επιταχύνετε, να ανακεφαλαιώσετε γρήγορα για να έρθει η επίτροπος. Έχουμε την τροπολογία 32 και εκεί περιμένουμε τη γνώμη σας στα μέλη της Επιτροπής. Θα είμαι σύντομος λοιπόν για την τροπολογία 20 ένας, ε, ένας από τους πίνακες αναφέρεται ε, στην συλλογική κατανάλωση κλπ. Αυτό καλύπτεται λόγω του, της ε, τροπολογίας που σχετίζεται. Έρχομαι λοιπόν στην 32. Το θύμα είναι ποιος είναι ο ορισμός της εστίασης του catering ε, για τις ε, στατιστικές στο ισοζύγιο πληρωμών και στους δορυφορικούς λογαριασμούς. Η εστίαση μπορεί να είναι σημαντική. Αν διατηρηθεί αυτή η τροπολογία θα ήταν καλύτερα να αναφερθούμε σε εστιατόρια και σε καφέ. Ε, τα προϊόντα που καταναλώνουν ε, οι τουρίστες από τα, υπηρεσίε υπηρεσίες που είναι τα εστιατόρια και τα καφέ και να αφαιρέσουμε τα, ε, τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ όπου αγοράζονται προϊόντα εστίασης. Σχετικά με την ε, τροπολογία 31 για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ε, έχουμε ε, έρευνες στις οικογένειες, δεν είναι ε, στοιχεία τα οποία συλλέγουμε από την, τις μονάδες στέγασης. Τότε τα δείγματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα και δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν καλά την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Επίτροπος είναι έτοιμη. Η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη θα έλθει εδώ στην Αθήνα.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 Λοιπόν. Είναι το κουδούνι της Επιτροπής αυτό ή της Επιτρόπου. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Σας ζητούμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που σας είχαμε αρχικά δώσει. Θα είμαστε ευγνώμονες αν μπορούσατε να μας μιλήσετε για 15 λεπτά περίπου μιλώντας για τον κανονισμό που καθιερώνει ένα πρόγραμμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυρία Μάιστιν, και να μας δώσετε μια γενική εικόνα του προγράμματος της Επιτροπής για τα ολοκληρωμένα θαλάσσια θέματα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας να έρθω να σας μιλήσω σήμερα εδώ. Όπως ξέρετε είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Είχα τη χαρά να έρθω και πέρσι τον Ιούνιο και να απαντήσω στα, στις ερωτήματα σας μετά από την έκθεση της κυρίας Μάσια για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αυτή η έκθεση είναι το τελευταίο παράδειγμα της συνεπούς υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια ναυτιλιακή πολιτική. Και θα σας πω ξεκάθαρα ότι έγινε πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά με αυτή την έκθεση, η οποία προσφέρει ένα συγκεκριμένο όραμα για την, ολοκληρωμένη θαλάσσια, για την ολοκλήρωση της θαλάσσιας πολιτικής με νέες οδούς που απλώνονται μπροστά μας, με προτεραιότητα την προώθηση της θαλάσσιας διάστασης της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Γι' αυτό θα θυμίσω όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και να αναφερθώ σύντομα σε κάποια από τα σημαντικά έργα που προβλέπονται για το 2011. Σχετικά με αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Το Σεπτέμβριο παραδώσαμε την ανακοίνωση ε, θαλάσσια γνώση 2020. Είμαστε πεπισμένοι ότι η θάλασσα προσφέρει τεράστιες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η εκμετάλλευσή τους και η αξιοποίησή του, ωστόσο απαιτούν περισσότερε γνώσει που θα επιτρέψουν τους επιστήμονε και τους μηχανικούς και του επιχειρηματίε Ευρωπαϊκή Ένωσης να προτείνουν νέε υπηρεσίε και νέα προϊόντα για την ανάπτυξη αυτή. Η πρότασή μα, για τη θαλάσσια γνώση έχει σκοπό να αξιοποιήσει πλήρω τα στοιχεία που υπάρχουν, που συγκεντρώνουν και διαθέτουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε πολλούς από τους άλλους στόχους που, έχουμε, ε, που έχουν τεθεί στην έκθεσή σας. Παραδείγματο χάρη και θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, θα μας βοηθεί να συναντιδρούμε πιο άμεσα στις ε, απρόβλεπτες ε, καταστροφές και στα λεπτά προβλήματα. Ενώ θα προσαρμοζόμαστε στην κλιματική αλλαγή με καλύτερες δυνατότητες ε, για μετρολογικές προβλέψεις. Αν περιορίσουμε την αβεβαιότητα για την αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 25% θα μπορέσουμε ε, να εξοικονομήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο προστατεύοντας τη Βενετία, το Λονδίνο και την Ολλανδία από τις άγριες θάλασσες και την άνοδο της στάθμης τους. Μόνο σε αυτούς τους τρεις τομείς, σε αυτές τις χώρες, η μείωση κατά 25% της αβεβαιότητας θα μας επιτρέψει να εξοικονομούμε 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η πρόταση λοιπόν έχει σκοπό να κάνει πιο αποτελεσματική, πιο προσβάσιμη τη συγκέντρωση στοιχείων και γνώσεων. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε ήταν η ολοκλήρωση της, ένα ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας παρακολούθησης με ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων. Ε, είναι μια πρωτοβουλία που την υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή και η Επιτροπή πριν από δύο εβδομάδες ε, ε, ε, εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα ώστε όλα τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν στοιχεία με έναν αποτελεσματικό και τρόπο. Θα συνεχίσουμε αυτή την ανταλλαγή στοιχείων το 2011 στο πλαίσιο δύο πιλωτικών προγραμμάτων και θα αρχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχετικό δικό χάρτη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει όλες τις δυνατότητες για την δημιουργία θέσεων εργασίας, μελετώντας πώς μπορούμε να να καταστήσουμε την κιανή ανάπτυξη μια πραγματικότητα. Αυτή η προπαρασκευαστική εργασία θα ενταχθεί σε μια ανακοίνωση για την κιανή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται για το 2012. Θα εξακολουθούμε να προωθούμε την αηφόρο ανάπτυξη τομέων όπως είναι η ενέργεια ή ο τουρισμός. Και με την, με την ανακοίνωσή μας για τον τουρισμό έχουμε τώρα ένα πολιτικό πλαίσιο για την προώθηση τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη και αν αξιοποιήσουμε, αν αξιοποιήσουμε και, αν, και με τη σωστή αξιοποίηση νέων ενεργειακών πηγών θα πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στις για ορισμένες ε, θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Με αυτό τον τρόπο θα αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία της ολοκληρωμένης προσέγγισής μας. Για το 2011 τι προβλέπετε. Ειδικό σχεδιασμός στον θαλάσσιο τομέα. Ευρωπαϊκή ζητήθηκε να, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προετοιμάσει μία πρόταση για δράση και αυτό κάναμε ώστε τα κράτη-μέλη να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του θαλάσσιου χώρου θα εστιαστούμε σε μια κοινή προσέγγιση για την θαλάσσια χωροταξία, ώστε να διευκολύνουμε την διασυνοριακή συνεργασία σε στενή επαφή με τα κράτη-μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οποιαδήποτε περαιτέρω δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πλαισιωθεί από ειδικέ πολιτικές, ενώ θα προωθείται η αρχή της επικουρικότητας. Αυτό είναι το μήνυμα που μας έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα προβεί σε μία αξιολόγηση επιπτώσεων για την ε, ε, χωροταξική ανάλυση των θαλασσίων χώρων και ε, θα θεσπίσουμε τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις για την προώθηση αυτού του θέματος με τη δική σας στενή συνεργασία. Επίσης, για του χρόνου προβλέπουμε την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για στις θαλάσσιες περιοχές, ξεκινώντας με την περιοχή του Ατλαντικού, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ατλαντικός έχει, προσφέρει μια σειρά από προκλήσεις, χαμηλές πυκνότητες πληκατοίκηση, <clears throat> αλλά ισχυρή άνεμη, υπαλλήρια και τα κύματα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα περιορίσουμε τον τρόπο αυτό της εκπομπές άνθρακα και θα περιορίσουμε την εξάρτησή μας από ορισμένους προμηθευτές. Ο Ατλαντικός είναι επίσης ένας ε, τομέας ο οποίος θα μας ε, επιτρέψει να συσφίξουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές ανταποκρινόμενοι στις επιταγές της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτές οι ε, οι προτάσεις οι οποίες είναι πολύ φιλόδοξες πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για εφαρμογή από το 2011 μέχρι το, 2013. Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, όπως μου ζητήθηκε, με φέρνει στο επίκεντρο των ρυθμίσεών μας, που είναι ένας κανονισμός ο οποίος θα καλύψει τη, τη, τις απομείνασες ε, δημοσιονομικές προοπτικές τίποτε δεν θα μας σταματήσει να προωθήσουμε την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών μας. Η χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ μετριοπαθής, κυρίως αν λάβουμε υπόψη ότι ο στόχος είναι τριπλός. Πρώτον, να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν το διερευνητικό τους έργο. Αυτό το έργο έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από προπαρασκευαστικές ενέργειες με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω και ε, διάφορες δυνατότητες για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής σε συνεργασία με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Δεύτερον, πρέπει να συμπληρώσει και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις μελλοντικέ χρηματοδοτήσεις των παράκτων περιοχών και των κρατών μελών. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να υπογραμμίσω. Δηλαδή, θα βοηθήσουμε τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από σε, περιοχές, σε περιφέρειες και κράτη-μέλη. Τρίτον, πρέπει να αναπτύξουμε συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και ε, πόρους οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εστιάζουμε λοιπόν, εστιαζόμαστε σε ορισμένες προτεραιότητες που θα εξασφαλίσουν ωφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν θα χρηματοδοτούμε τα προγράμματά μας, θα χρηματοδο... μόνο γενικά προγράμματα, αλλά μόνο προγράμματα που θα προσφέρουν ωφέλη σε όλους εμάς, ε, οργανισμούς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κλπ. Σας απευθύνω λοιπόν έκκληση κύριε Πρόεδρε, να δώσετε άμεση προτεραιότητα στην ε, διαδικασία έγκρισης αυτού του κανονισμού, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό το 2011. Ο ενθουσιασμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δεδομένος. Το σχέδιο ψηφίσματος με βάση την έκθεση Μάισνερ καλεί ζητά την γρήγορη θέσπιση του κανονισμού αν το κάνουμε αυτό θα δείξουμε ότι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι αυτή η πολιτική. Η Κομισιόν προσβλέπει στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Έχουμε ήδη δει τι μπορεί να κάνει αυτή η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Με την κατάλληλη υποστήριξη θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, είμαι πεπισμένη ότι με την υποστήριξή σας το 2011 θα είναι ένα εξαιρετικό έτος για την ε, πολιτική μας. Προσβλέποντας ε, προς το μέλλον, όλες, ε, όλα τα τμήματα της Επιτροπής εργάζονται για τις δημοσιονομικές προπτικές που θα μας οδηγήσουν στο 2020. Προσπαθούμε λοιπόν να εντάξουμε την θαλάσσια διάσταση σε όλα τα σχέδια χρηματοδότησης μετά το 2013. Αυτό είναι σωστό, διότι όλες οι θαλάσσιες πολιτικές μπαίνουν στο κεντρικό πρόγραμμά μας για τη μελλοντική ευημερία και ανάπτυξη. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ορίμασε και χρήζει της υποστήριξής σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, για αυτή την εισήγηση. Θα ήθελα να εγγραφούν στον κατάλογο όλοι οι ομιλητές. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει το λόγο του ονόματος του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή μας. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι μια νέα πολιτική. Εγκαινιάστηκε μόλις το 2007 αλλά προχωράει με έναν δυναμικό βηματισμό και αυτό είναι αναμφισβήτητο και το επιβεβαιώνει άλλωστε και η σημερινή σας παρουσία και παρέμβαση εδώ. Ε, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι αναμφισβήτητα μια φιλόδοξη πολιτική. Όλοι μας αναρωτιόμαστε όλοι όμως εάν είναι και ανάλογα ρεαλιστική. Διότι οι στόχοι είναι πολλοί και κυρίως ο στόχος του συντονισμού επιμέρους τομέων που σχετίζονται με τη θάλασσα, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την αλία είναι εύκολο να λέγεται και να επιδιώκει το συντονισμός, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε όταν πάμε να τον επιδιώξουμε και να τον εφαρμόσουμε. Ταυτόχρονα έχετε τρει στόχου, τη θαλάσσια διακυβέρνηση, τη θαλάσσια επιτήρηση, τη θαλάσσια χωροταξία. Θα ήθελα να ρωτήσω σε, μια, σε ένα πρώτο στάδιο αν αυτοί οι τρει στόχοι του αναπτύσσετε παράλληλα ή αν έχετε θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες τι από αυτούς τους τρεις στόχους, ποιος από αυτούς είναι μπροστά και ποιος ακολουθεί, αν υπάρχει συγκεκριμένο επίσης ε, χρονοδιάγραμμα. Έρχεται βεβαίως εδώ και ανακύπτει το κέριο ερώτημα της χρηματοδότησης. Μιλήσατε για τα 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2013. Αναμφισβήτητα είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ε, μεγάλο για να στηρίξει μια τόσο φιλόδοξη πολιτική. Και προκύπτουν και ορισμένα ερωτήματα. Ε, κυρία Επίτροπε, εδώ. Παραδείγματο χάρη, μας μιλήσατε για την ανάγκη να προχωρήσει η θαλάσσια χωροταξία. Δεν, ε, δεν γνωρίζω και δεν το αναφέρατε εάν ε, η εξέλιξη σε αυτό το σχέδιο σχετίζεται και μέχρι ποιο βαθμό από την εφαρμογή από όλα τα παράκτια κράτη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 διότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να προχωρήσει σε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με κράτη τα οποία δεν έχουν ως βάση αναφοράς τους τη διεθνή αυτή σύμβαση. Και θα ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Για τη θαλάσσια επιτήρηση. Άκουσα με προσοχή ε, τα σχέδιά σας, τα οποία υποστηρίζουμε όλοι. Ε, δεν ε, έχω αντιληφθεί αν μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο ε, προγραμματισμό που κάνετε έχετε εντάξει και την ΕΜΣΑ και τι ρόλο έχει η ΕΜΣΑ μέσα στην ε, προώθηση της θαλάσσιας επιτήρησης. Κυρία Επίτροπε, δεν θέλω να μακρηγορήσω πέραν ε, του λογικού. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ε, όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά αυτή η Επιτροπή στηρίζουν τις προσπάθειές σας. Αλλά ε, αυτό θα το κάνουμε με μεγάλη προσοχή και πάντως από πλευρά μα θα επιχειρήσουμε ότι ο κανονισμό αυτό, το σχέδιο κανονισμού που έχετε ήδη παρουσιάσει, να προχωρήσει με του ρυθμού που έχουμε δεσμευτεί, δηλαδή μέσα στο 2011. Thank you. Mr. Ευχαριστούμε. Κύριε Κουμουτσάκο, ο κύριος Δανέλη Κύριε... Ο κύριος Δανέλης από τους Σοσιαλιστές. Είμαστε ξανά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ καθώς επίσης και την φιλόδοξη ατζέντα σας για τα ζητήματα της εφαρμογής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Ε, η αντίληψη δική σας νομίζω ότι στα περισσότερα σημεία αποτελεί μια συναντήληψη με τον προβληματισμό και τις αγωνίες μας για την εφαρμογή της περίφημης ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, ζητήματα που για την Επιτροπή μας είναι κορυφαίας σημασίας μιας και όλοι έχουμε αντίληψη ότι στο σύνολό τους σχεδόν οι πολιτισμοί των λαών της Ευρώπης διαχρονικά με στο πέρασμα των αιώνων βασίστηκαν με καθοριστικό τρόπο στη θάλασσα, στη σχέση τους με τη θάλασσα. Ε, και νομίζω ότι όλοι βιώνουμε και όλο και περισσότερο με την αύξηση των πιέσεων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης βιώνουμε τα προβλήματα ε, οργάνωσης των διαφορετικών χρήσεων που όλες έχουν αντικείμενο την θάλασσα είτε τις παράκτιες περιοχές ε, και βεβαίως ε, κάποιες φορές οι συγκρούσεις των χρήσεων ε, δημιουργούν τεράστια προβλήματα με κόστος κοινωνικό και οικονομικό. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η θαλάσσια χροταξία είναι μίζωνος σημασία στόχος άλλο τόσο βεβαίως είναι και εξαιρετικά δύσκολο ε, να εφαρμοστεί και να είναι αποδεκτό από το σύνολο των ε, χωρών μελών. Ε, έτσι λοιπόν όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια, διασυνοριακή οργάνωση της θαλάσσιας... του θαλάσσιου χωροκρατικού σχεδιασμού. ένα μείζονο σημασίας επίσης θέμα για μία από τις δραστηριότητες, ίσως μία από τις σημαντικότερες που αφορούν στην ε, θάλασσα είναι η ναυτιλία βεβαίως και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία είναι προτεραιότητας για όλους μας για να μπορέσει να ε, λειτουργεί ο κλάδος και να ευημερεί όχι μονάχα στην Ένωση θα πρέπει να πετύχουμε ένα ψηλό επίπεδο ε, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία. Ε, νομίζω ότι στις μέρες μας υπάρχει ένας επιπλέον ε, φόβος για την ε, συνέχεια της αδιατάραχτης λειτουργίας της ναυτιλίας που έχει να κάνει με την πειρατεία. Βεβαίως, όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς σε ευρωπαϊκό πλαίσιο όμως νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες στα πλαίσια του ΟΗΕ να υπάρξει μια άλλου είδους αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος που γίνεται όλο και μεγαλύτερο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί βεβαίως μονάχα ε, στρατιωτικά επιχειρησιακά. Ε, έτσι θα ήθελα να μάθω αν μέσα στην ατζέντα σας υπάρχει κάτι για την αντιμετώπιση της πειρατείας και τη λήψη πρωτοβουλειών από μέρους σας. Ε, τέλος θέλω να ε, μας πείτε πώς βλέπετε την ενεργοποίηση, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, πώς ενισχύει τη θαλάσσια διακυβέρνηση, πώς ενεργοποιούνται ε, και πώς ουσιαστικά συμμετέχουν και μάλιστα με μόνιμη ένταξη στις δομές όλοι οι εμπλεκόμενοι, περιφερειακές και εθνικές βεβαίως αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ξέρω ότι έπρεπε να βρείτε χρόνο για να μας υποβάλλετε αυτή την έκθεση σήμερα. Εγώ αναγνωρίζω τη σημασία του θέματος. Χρειαζόμαστε μια γενική πολιτική, μια κεντρική πολιτική, mainstreaming αυτής της πολιτικής, την οποία ακόμα δεν έχουμε επιτύχει. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αρχίσουμε με την χρηματοδότηση και σε ποιο σημείο βρίσκεστε ως προς τη χρηματοδότηση θα πρέπει να την θέσουμε σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν για το 2011. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να αναθεωρήσουμε τη θαλάσσια πολιτική και να την χρηματοδοτήσουμε συνάμα. Από πού θα αρχίσετε, τι ιεράρχηση θα κάνετε, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει αυτή η πολιτική ένα γενικό ευεργέτημα για τους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ζητήματος. Ως προς την ανταλλαγή δεδομένων, νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί η θάλασσα ενέχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό Δηλαδή έχουμε 15.000 ε, προϊόντα τα οποία την χάνουν έρευνας. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και γαλάζιες θέσεις απασχόλησης για την διερεύνηση της θάλασσας. Επίσης, ως προς τις πρώτες ύλες ε, θα πρέπει να προωθηθεί μια συζήτηση για τους θαλάσσιους πόρους. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε επιστημονικά προγράμματα για να προωθήσουμε την ολοκληρωμένη πολιτική. Το θέμα της επαγρύπνησης και της ασφάλειας επίσης είναι ύψης της σημασίας. Και επ' αυτού συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες ότι πρόκειται δηλαδή για ένα γενικότερο θέμα διασάφησης. Πού έχουμε αρμοδιότητες και πού όχι, γιατί υπάρχει μία σύγχυση σε σχέση με τις αρμοδιότητές μας, ιδιαίτερα γύρω από τη Μεσόγειο. Πώς μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτόν τον προγραμματισμό. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα των θαλάσσιων πόρων και επίσης να αντιμετωπίσουμε και θέματα της ανοιχτής θάλασσας ως προς τα ατυχήματα, τι μπορούν να μας μάθουν αυτά τα ατυχήματα στην ανοιχτή θάλασσα και πώς ε, μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Θα πρέπει να προβάλλουμε μία στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική ναυπηγικής. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να προβάλλουμε μία τέτοια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να προωθηθεί αυτό το ζήτημα, διότι θα μπορούσε να οδηγήσει και σε νέες θέσει εργασίας. Ο κύριος Βαντάλεν. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, κύριε Επίτροπε, σχετικά με την δική μου ομάδα και αυτή την πρωτοβουλία νομίζουμε ότι είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αναμένουμε. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για μας, η επικουρικότητα πρώτον και το θέμα της βελτίωσης των παροχών των υπηρεσιών ως προς το περιβάλλον, κυρίως των θαλασσίων μεταφορών. Αναπτύσσοντας ορισμένα ε, τμήματα, ορισμένες δραστηριότητες όπως γίνεται στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο σημεία. Βεβαίως ε, δεν είμαι πλήρως ενήμερος ε, για το χαρτοφυλάκιο και πώς το μοιράζεστε το χαρτοφυλάκιο με τον κύριο Καλάς. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω πώς εξελίσσεται η έρευνα της Κομισιόν σχετικά με το επίπεδο του 0,1% ε, θείου στα καύσιμα των πλοίων ε, στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό ισχύει για τη Βαλτική, για τη Βόρεια Θάλασσα και για άλλες περιοχές, αλλά πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι μπορεί να υπάρχει σημαντική εκπομπή, εκπομπές άνθρακα και βεβαίως αυτό μπορεί ε, να θέσει ε, θέματα ανταγωνισμού, διαταραχής του ανταγωνισμού. Δεύτερον, οι διαπραγματεύσεις για ένα σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπής δεν είναι ακόμα ένα σύστημα πάρα πολύ χρήσιμο. Πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα αποτελέσματα στον Διεθνή Ναυτοριακό Οργανισμό. Δεν μπόρεσε ο οργανισμός να εξαγάγει συμπεράσματα, αλλά ε, από ό,τι ξέρω θα ήθελα ε, να μου πείτε εσείς ποια είναι η θέση σας, τι ξέρετε σε σχέση με τέτοια συστήματα πολύ καλά. Τέλος. Τέλος, ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας συναντήσετε. Μιλάμε για... τις θαλάσσιες μεταφορές. Όταν όμως φτάνουμε στο πρόβλημα των εκπομπών, δεν υπάρχουν διατάξεις για το πώς στην ανοιχτή θάλασσα μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις εκπομπές. Έχουμε ε, εγκαταστάσεις ε, καύσης χωρίς φίλτρα και τα βαρέα έλαια που δεν χρησιμοποιούνται, που είναι απόβλητα και που θα έπρεπε να καθαρίζονται πρώτα αλλά δυστυχώς απορρίπτονται στη θάλασσα. Και θεωρούμε ότι το θέμα έχει λήξει. Οι μεταφορές στην ανοιχτή θάλασσα είναι ε, κάτι που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για το περιβάλλον. το κόστος της μεταφοράς όταν πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πλοίο δεν είναι ενδεχομένως πάρα πολύ μεγάλο. Και όμως αυτά τα πλοία αρνούνται να κάνουν οτιδήποτε, οτιδήποτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Μόνο στη θάλασσα γίνονται αποδοκτά αυτά τα συστήματα καύσης χωρίς καθαρισμό. Για δύο λόγια, δύο λεπτά ο κύριος Ρίκελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε να μας συναντήσει και θα είμαι πολύ σύντομος. Ως εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμού για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Όταν βλέπουμε όμως τον όγκο που αποτελεί η θάλασσα ε, και οι παράκτης περιοχές και βλέπουμε τα ποσά που διαθέτεται, 50 εκατομμύρια μόνο, προκύπτουν ερωτήματα για το, την έκταση του προγράμματος, για την έκταση των δράσεων και την πάρα πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση που προβλέπεται για αυτά. Ερωτώ λοιπόν, πώς προβλέπετε πέρα από τον καθορισμό των προγραμμάτων που μας δώσατε, πώς Πώς βλέπετε αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε σχέση με τον προϋπολογισμό της. Θα περιοριστούμε στις μελέτες ή θα υπάρξει δυνατότητα να συγκεντρώσουμε τις μελέτες που εκπονούνται από τα κράτη-μέρη, θα προβλεφθούν άμεσες δράσεις και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρησιακών δράσεων μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ διαφόρων χωρών. Διότι βλέποντας το, το χαμηλό επίπεδο του προπολογισμού σας, διερωτώμαστε πώς θα τα υλοποιήσετε όλα αυτά που μας ανακοινώσατε. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που παρευρίσκεστε εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική ανησυχία εξ ονόματος όλων για το πώς θα έχει η κατανομή των 50 εκατομμυρίων και πώς θα γίνει ένας επιμερισμός χρηματοδοτήσεων. Και αυτό γενικότερα για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να μιλήσουμε για ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αλλά να ξέρουμε ε, κατά πόσο στηρίζει και μία κοινή και την κοινή αλλιευτική πολιτική. Επίσης, ο τομέας της ναυπηγικής γνωρίζει μεγάλο ανταγωνισμό από την νοτιοανατολική Ασία και βεβαίως και οι αλλοιείς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ως προς την ασφάλειά τους. Υπάρχει και το θέμα της πειρατείας, της καινοτομίας, του συντονισμού. Αυτά τα είπε και ένας άλλος βουλευτής από τους σοσιαλιστές. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε αυτή την πορεία κατά τα επόμενα χρόνια. Γιατί βεβαίως οι μελέτες θα μας δώσουν καλύτερα στοιχεία. Αλλά τι προβλέπετε για τα δύο επόμενα χρόνια. Θα υποστηρίξουμε την κοινή αλλιευτική πολιτική. Τι θα γίνει με τις συμφωνίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τις συμβάσεις. Τι θα γίνει με το τομέα της ναυπήκης. Τι θα γίνει με τις παράκτιες περιοχές όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Θα ήθελα να γίνει μία ιεράρχηση, να γνωρίζουμε μία σαφή πολιτική. Γιατί θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο εσείς οι Επίτροποι μεταξύ σας έχετε προβλέψει ένα συντονισμό ως προς την κατανομή αυτών των κονδυλίων. Μιλάμε για δύο, τρία, τέσσερα σχέδια, μιλάμε για εξυγχρονισμό, για απασχολησιμότητα. Θα ήθελα να μας πείτε σε ποια ιεράρχηση έχετε προβεί και κατά πόσο υπάρχουν, υπάρχει συντονισμός μεταξύ επιτρόπων. Θα ήθελα να μας πείτε πώς κινείστε ως προς αυτό τον κοινό συντονισμό μεταξύ σας. Και εγώ θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις, κυρία Επίτροπη. Σε σχέση με την αυπηγική και θα ήθελα να μιλήσω και για τον παραπλησμό των ε, πλοίων. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα κάνουμε με τη βιομηχανία ship breaking, με τον παροπλισμό των ε, πλοίων. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και από άλλα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα από την Ασία. Επίσης, τι θα γίνει με τα κοντέινερ θα θυμόσαστε ότι πολλά εμπορευματοκιβώτια έπεφταν από τα πλοία. Και αυτό αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την αυσιπλοεία γενικότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Μην ξεχνάμε ότι 20.000 εμπορευματοκιβώτια χάνονται κάθε χρόνο. Αυτό να το δούμε μαζί με την διάλυση των πλοίων. Πώς θα προβάλλουμε αυτή την πολιτική. Μπορούμε κάτι να κάνουμε και με τη γραφειοκρατία την οποία διαιωνίζουν τα κράτη-μέλη. Ακόμα και ενδοκινοτικά. Γιατί αυτό στην ουσία συρρυκνώνει την ανάπτυξη. Δεν πρέπει να ξεχνάτε τι εφιάλτες ε, ε, γνωρίζει ο τομέας της ε, ναυπηγικής και της ναυπήγησης, ιδιαίτερα ως προς τη μεταφορά φορτίων από τον ένα λιμένα στον άλλο. Ας καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία των τελωνίων, των ελέγχων, όλα αυτά θα βοηθούσαν ιδιαίτερα την θαλάσσια πολιτική. Και έχετε το λόγο, κυρία Επίτροπε, για τα υπόλοιπα δέκα λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που πήραν το λόγο για τις παρατηρήσεις τους, παρατηρήσεις που εκφράζουν και τις δικές μου σκέψεις, διότι πρόκειται για μια νέα πολιτική, όπως είπατε και εσείς, και πρέπει με προσοχή να δούμε ποιος θα είναι ο ρελιστικός τρόπος για να προχωρήσουμε. Πρώτος μας στόχος ήταν να έχουμε μερικές επαφές με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό Είπαμε πολλά για τα θέματα, τα κυβερνητικά και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ελπίζω ότι θα έχουμε ένα δίκτυο με τα κράτη-μέλη, με μερικούς εκπροσώπους ε, της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε σημεία επαφής σε όλα τα κράτη-μέλη, το, ε, το δουλεύουμε γι' αυτό, ε, δεν χρειάζονται χρήματα για τέτοιο ε, θέμα, για τέτοιο δίκτυο, δεν χρειάζεται χρηματοδότηση, αλλά αν πείσουμε τα άτομα αυτά ότι θα υπάρξει προστιθέμενη αξία, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε αυτό το δίκτυο με τις κυβερνήσεις και να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αυτά τα θέματα αγριοφυκρατίας που ανέφερε ο Πρόεδρος. Έχουμε μετά αυτούς τους τρεις πυλώνες της πολιτικής μας. Ε, θαλάσσια γνώση, θαλάσσια επιτήρηση και ειδικό προγραμματισμός θαλάσσιος. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο καθένα Τι γνώση και θα ήθελα να εξηγήσω λογικά με ορισμένα παραδείγματα. Τι, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις συνδέσεις ανάμεσα σε όλα τα έργα, σε όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη γνώση και τη θάλασσα. Για του χρόνου, παραδείγματο χάρη, έχω συνεργαστεί με την, με, τον Επίτροπο για με την Επίτροπο για την Έρευνα, την κυρία Κουίν, και αποφασίσαμε ε, να θεσπίσουμε ένα ε, πρόγραμμα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς του αύριο. 45 ε, εκατομμύρια. Έχω λοιπόν συνεργασία με την άλλη Επίτροπο, αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν είναι το μόνο, το μόνο θέμα που έχουμε χρηματοδότηση για θαλάσσια έρευνα. Έχουμε πάρα πολλά κονδύλια για την έρευνα την θαλάσσια. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στη χρηματοδότηση πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι χρειαζόμαστε αυτά τα 50 εκατομμύρια για να δημιουργήσουμε τις συνδέσεις ανάμεσα σε τομείς που έχουν πολλά εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια δεν είναι το, το ποσό που αναφέρεται σε αυτές τις δράσεις. Τα 50 εκατομμύρια περιορισμένο κονδύλιο θα μας επιτρέψει να έχουμε ε, τις ε, συνδέσεις ε, ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα και έργα. Με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτή η θαλάσσια έρευνα είναι ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε 41 εκατομμύρια για το επόμενο έτος από την χρηματοδότηση για έρευνα για θαλάσσιες δράσεις, αλλά έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για την έρευνα γενικά. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε. Και ποιο είναι το πρόβλημά μας εδώ. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε διαπιστώσει από τη δική μας άποψη και αναφέρομαι τώρα στην αυπήγηση. Στην αυπηγική έχουμε πολλά προγράμματα ερευνητικά σχετικά με τα καθαρά πλοία, σχετικά με την, την καινοτομία στην, στον αυπηγικό τομέα, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο στάδιο της εμπορικοποίησης, εμπορευματοποίησης. Πρέπει να πείσουμε τις υπηρεσίες της Κομισιό να δώσουν τα κονδύλια στα προγράμματα τα οποία συνδέουν τα, ερευνητικά προγράμματα και τα προγράμματα καινοτομία με την ναυπηγική δραστηριότητα και αυτό είναι κάτι ε, που ε, θα κάνουμε με αυτά τα κονδύλια. Έχουμε το πρόγραμμα και χρειαζόμαστε τα κονδύλια για να συνδέσουμε αυτά τα προγράμματα. Βεβαίως η ναυπηγική, τα ναυπηγεία, η διάλυση των πλοίων, η ασφάλεια των πλοίων. Αυτή δεν είναι αρμοδιότητά μου, αλλά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην υπηρεσία μου και και τις του κυρίου Κάλλας. Και παραδείγματο χάρη η ΕΜΣΑ θα λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα επιτήρησης. Θα σας εξηγήσω τι θα γίνει για να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Κουματσάκος. Η ΕΜΣΑ θα έχει τις επαφές της. Δεν πρόκειται αυτόν τον τομέα. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε θα προσπαθήσουμε ε, ε, να, έχουμε όλα τα στοιχεία από όλη την έρευνα για, με την, ε, υπηρεσία ασφάλειας για να προσπαθήσουμε να η ΕΜΣΑ θα μας δώσει κάτι διότι παίρνουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη, από τις εθνικές αρχές, από τις στρατιωτικές αρχές. Πρόκειται να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία ούτω ώστε όλα αυτά να μπορέσουμε να τα εξασφαλίσουμε για να έχουμε τα προγράμματα ασφαλείας, διότι στόχος μας ε, σχετικά με την επιτήρηση, την επίβλεψη, δεν είναι να, την υπηρεσία αυτή ασφαλείας ε, να την αντικαταστήσουμε, αλλά να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία, ούτω ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους. Ε, με αυτά τα 50 εκατομμύρια που είναι ένα μικρό ε, ποσό είναι να έχουμε ένα ε, πιλωτικό πρόγραμμα, πραντό χάρη για την Μεσόγειο που κάναμε πολύ καλή δουλειά για να δώσουμε τα στοιχεία αυτά σε όλους. Αυτή ήταν η προστιθέμενη αξία. Να πείσουμε τους άλλους ότι ε, θα γίνουν αυτά. Επίσης έχουμε εργαστεί με τον κύριο Ποτόκιν, διότι ε, για την, ε, με τον ειδικό προγραμματισμό του, ώστε με τον κύριο Ποτόκιν, τον Επίτροπο για το Περιβάλλον, να ασχοληθούμε με την διαχείριση των παρακτήων περιοχών και θα έχουμε μια μελέτη αντικτύπου για αυτές τις δράσεις. Θα δημιουργήσουμε συνέργειες και θα είναι ευκολότερο μετά για την Επιτροπή να αντιδράσει. Σχετικά με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τις εκπομπές, ε, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ε, σχετικά με τις εκπομπές αλλά όχι για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, αλλά του NO. Μιλάω στην Επιτροπή Μεταφορών. Το ξέχασα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον αυτιλιακό οργανισμό για να βρούμε ένα consensus, ε, διότι η θέση της Επιτροπής εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί να έχει την δική της, ε, τη δική της νομοθεσία, μόνο νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με την νομοθεσία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, διότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ο θαλάσσιος, ο ναυτιλιακός τομέας δεν θα είναι ανταγωνιστικός. Ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτές τις εκπομπές, δηλαδή τι θα κάνουμε χρειαζόμαστε θαλάσσιες μεταφορές ε, καθαρές, αλλά οι θαλάσσιες μεταφορές ακόμα και τώρα είναι πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τους άλλα μέσα μεταφοράς, ε, από ότι τις χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων, ε, φορτίων. Ε, βήμα προς βήμα προχωρούμε με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Αυτά μπορώ να σας πω. Σχετικά με τη γραφειοκρατία και σχετικά με τον τομέα τον ναυτιλιακό και ναυπηγικό. Αν έχετε ένα φορτίο και πρέπει να τον μεταφέρετε διοδικής ε, μεταφοράς είναι ευκολότερα. Η ΕΜΣΑ, η Υπηρεσία Ασφαλείας και οι υπηρεσίες του κυρίου Κάλλας έχουν θεσπίσει μια διαδικασία ούτω ώστε να υπάρχει ένας τομέας εσωτερικής αγοράς ε, για ε, την ακτοπλοεία. Και σχετικά με την πειρατεία, να προσθέσω κάτι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Κύριε Δανέλη, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Είχαμε την Αταλάντα, την επιχείρηση Αταλάντα με το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά έχουμε απαγωγές ευξημένε, έχουμε επίσης ευξημένε απαιτήσει για αποζημιώσεις για να ελευθερωθούν αυτά τα άτομα τα οποία είναι θύματα της ε, πειρατείας. Πρέπει να κάνουμε κάτι και η Λέιδη Άστον η οποία είναι αρμόδια πρόκειται να ασχοληθεί με το θέμα. Ε, σχετικά με την χρηματοδότηση Νομίζω ότι το ποσό αυτό είναι μικρό, αλλά αυτό που θέλω να κατανοήσετε είναι ότι το κονδύλιο αυτό δεν το χρησιμοποιήσουμε απλώς για να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Θα χρησιμοποιήσουμε το κονδύλιο απλώς για μελέτες και για πιλωτικά προγράμματα για να δημιουργήσουμε συνδέσεις ανάμεσα σε προγράμματα που υπάρχουν ήδη και για να προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε ορισμένα πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα μας δώσουν μια προστιθέμενη αξία στην πολιτική μας. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ μικρό κονδύλι αν το σκεφτείτε έτσι, αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι χρειαζόμαστε πράγματι την υποστήριξή σας, διότι δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θα μας δώσει ακόμη και αυτό το μικρό κονδύλιο λόγω της κρίσης, λόγω ε, της ε, γενικών τάσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα, μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να είμαστε συγκεκριμένοι ακόμα ε, και να ξοδέψουμε ακόμα και το τελευταίο ευρώ για να πείσουμε όλους ότι έχουμε ένα πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα. Ξέχασα να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Αυτό που ήθελα να σας πω κύριε Κουμουτσάκο είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την αξιολόγηση επιπτώσεων για την ε, διαχείριση των ακτών και των θαλάσσιων χώρων για να δημιουργήσουμε αυτές τις συνδέσεις. Κανένας που θα συνεργαστεί μαζί μας δεν έχει υποχρέωση να επικυρώσει τη σύμβαση, την οποία όμως την έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα προκύπτει μόνο με τις τρίτες χώρες. Και αυτό το είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη διεύρυνση και την πολιτική καλή γειτονία. Πρόκειται λοιπόν για πολιτικό ζήτημα και θα λάβουμε τη σχετική απόφαση σε ό,τι αφορά δηλαδή τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας αύριο στο Σώμα των Επιτρόπων. Thank you very much again. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε να μας συναντήσετε και όπως ξέρετε υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από πλευράς της Επιτροπής μας για τις προτάσεις που αφορούν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναπτύξουμε το θαλάσσιο τομέα μας, τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε που μας αφιερώσατε το χρόνο σας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Τώρα θα έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών.